Κυρίες και κύριοι, μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο μπορούμε να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Η καθυστέρηση και το ακαδημαϊκό τέταρτο ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα η απογευματινή συνεδρίαση. Γι' αυτό επιτρέψαμε αυτή την καθυστέρηση το ακαδημαϊκό τέταρτο. Είναι εξαιρετική η σημασία η απογευματινή μας συνεδρίαση, γιατί έχουμε έναν υψηλό προσκεκλημένο. Έναν άνθρωπο που έκανε πάρα πολλά για μας και εξακολουθεί να προσφέρει πολλά στην Ήπεθρο και στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και μάλιστα πολύ συχνά το έκανε να το να σε δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό και όταν περνούμε και εμείς δυσκολίες και έχουμε αντίξωες συνθήκες, θυμόμαστε τον Επίτροπο Φίσλερ, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας σήμερα. Επιτέλεσε πολύ σημαντικό έργο ως Επίτροπος και είχα την ευκαιρία να τον δω και να το θαυμάσω από κοντά. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσλερ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας, που ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε... Θα θέλαμε να μας παρουσιάσετε τις απόψεις σας για πολλά σημαντικά και δύσκολα πράγματα που μας ταλανίζουν και στις χώρες μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που αφορούν κυρίως την αγροτική ανάπτυξη, την Ήπεθρο γιατί η κοινή γεωρική πολιτική αποκτά όλο και περισσότερες ε, εξωτερικές διαστάσεις, επηρεάζεται όλο και περισσότερο από εξωτερικούς παράγοντες. Ε, έχουμε τη συζήτηση για το TTIP, τη νέα εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ δύσκολα θέματα και το πρωί είχαμε πολύ σημαντική και σφοδρή συζήτηση για την πολύ δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να, να ακούσουμε και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά. Έχουμε τώρα τον κύριο Φίσλερ που είναι ο πρόεδρο τη Επιστημονική Οργανωτική επιτροπή τη ΕΞΠΟ του Μιλάνου για το 2015. Κύριε Φίσλερ, έχετε επιρροή, επηρεάζετε κάποια ουσιαστικά θέματα της ΕΞΠΟ Και ο προκάτοχός μου, ο κύριος Δεκάστρο, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την έξπο του Μιλάνου για το 2015. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την παρουσίασή σας αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία για πολύ πιο εκτενή συζήτηση για τις γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κοινή γεωρική πολιτική. Έχετε το λόγο λοιπόν τώρα, κύριε Φίσλερ, παρακαλώ. Chairman, I can assure you it will not Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα είμαι πάρα πολύ ακαδημαϊκός αυτά τα οποία θα σας πω, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη. Σε 177 ημέρες από σήμερα το Expo Μιλάνο 15 θα ανοίξει τις πόρτες της. Μια μοναδική ευκαιρία για την Ευρώπη να αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντός μας, πώς να παράγουμε με ασφαλή τρόπο και αηφόρο τρόπο επαρκή τρόφιμα για όλη την ανθρωπότητα. Είμαι πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής που ξεκίνησε τον μήνα Μάρτιο. Περιλαμβάνει 11 εμπειρογνώμονες από το σύνολο της Ευρώπης και πέραν αυτής με στόχο να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα που θα χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της Expo Μιλάνο 2015. Θέλουμε να συνεισφέρουμε στην συνέχεια, στην κληρονομιά της Expo, αναπτύσσοντας επιστημονικές θέσεις για τη διασφάλιση της προμήθειας των τροφίμων. 147 χώρες, πάρα πολλές διεθνείς οργανώσεις, ε, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών θα πάρουν μέρος σε αυτήν την μεγάλη διεθνή έκθεση και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή και να καθορίσει τον ρόλο της σαν βασικός παίκτη στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων. Τίτλος είναι «Τροφή για τον πλανήτη και ενέργεια για τη ζωή». Είναι κάτι το οποίο διασταυρώνεται με πάρα πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές στην ανάπτυξη, στην ασφάλεια των τροφίμων, στο περιβάλλον, στην έρευνα, στην καινοτομία και τη βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην χάσει την ευκαιρία αυτή και να προσφέρει στην συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων και την αηφορία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο να δείξουμε ε, την εξαιρετική ποιότητα του ευρωπαϊκού ε, τροφιμικού τομέα στο Μιλάνο, όπως επίσης και το υψηλό επίπεδο της έρευνας στον ίδιο τομέα, αλλά να υπάρξει και καρποφόρα συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους και να προσκαλέσουμε την διεθνή την επιστημονική κοινότητα να εμπλακεί πλήρως στον διάλογο. Ένα θέμα το οποίο ξεκαθάρισε από την αρχή είναι η συμμετοχή. Η έρευνα και η καινοτομία είναι κεντρικά σημεία αντιμετώπισης των πιέσεων στο διεθνές τροφιμικό σύστημα και κάλυψης των αναγκών ε, στον τομέα των ζωικών πρωτεϊνών μια ζήτηση η οποία αυξάνεται συνεχώς λόγω της αύξησης του πληθυσμού. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε επίσης και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο εσωτερικό της γεωργικής παραγωγής. Όμως ε, οι περιορισμοί οι οποίοι τίθενται από τις κλιματολογικές αλλαγές, η έλλειψη των υδάτων όπως επίσης και η έλλειψη γεών και η χρήση γεών για μη γεωργικές ε, στόχους δημιουργούν προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι μόνο μέσω της καινοτομίας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ε, να ε, επιτρέψει να υπάρξουν περισσότερες αποδόσεις αλλά και με αηφορία. Γι' αυτούς τους λόγους λοιπόν ο λόγος ύπαρξης της Επιτροπής της Επιστημονικής είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει έναν δραστήριο ρόλο στα πλαίσια της ΕΞΠΟ 2015, να προωθήσει τις ιδέες της και να συνεισφέρει ε, στην διεθνή συζήτηση. Τον προηγούμενο μήνα η Επιτροπή Διοικητική ε, συζήτησε ένα πρώτο έγγραφο για τις μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στα τρόφιμα. Το έγγραφο αυτό έχει σαν βασικό στόχο να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους η ευρωπαϊκή έρευνα μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία. Θα είναι η βάση για τη συζήτηση με τους εμπλεκομένους και με το κοινό. Κατά τη διάρκεια της ΕΞΠΟ 2015 θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε όλες οι πλευρές ε, της ασφάλειας των τροφίμων να καλύπτονται και θα υπάρξει χώρος και χρόνος για συζητήσεις, διαβουλεύσεις και ανταλλαγές πρακτικών εμπειριών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να συμβάλλουμε στην κληρονομιά της ΕΞΠΟ. Να μου επιτρέψετε λίγο να σας πω το τι ακριβώς ε, θα μας απασχολήσει. Ε, τα προβλήματα της ασφάλειας των τροφίμων. Εδώ οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι απαιτούνται νέες γνώσεις σε επτά τομείς. Πρώτος τομέας, βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσω της διατροφής. Πώς μπορούμε να τρώμε αηφόρα και με υγιεινό τρόπο. Δεύτερον, να καταστήσουμε την τροφιμική αλυσίδα πιο αποτελεσματική, να μην υπάρχουν απώλειες, να βελτιωθεί η ποιότητα των τροφίμων να διαχειριστούμε τα τρόφιμα σε ένα ολοένα αυξανόμενο σφαιρικό σύστημα, να αυξήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα των τροφίμων, να διαχειριστούμε την γη ε, για πολλαπλούς στόχους προσαρμογής στις ανάγκες της φύσης κτλ. Και τέλος, αύξηση των αποδόσεων με αηφορία δηλαδή στην ουσία αυτό που θα ονομάζαμε αηφόρος εντατικοποίηση. Πολλά από τα θέματα αυτά είναι από τη φύση τους διεπιστημονικά, πολυτομεακά και δημιουργούν και θέματα σε επίπεδο πολιτισμικό. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λόγους να παρέμβει στον τομέα αυτό μέσω και του συντονισμού και της ευθυγράμμισης της έρευνας αναλαμβάνοντας την διεθνή ηγετική θέση στον τομέα της έρευνας για τα τρόφιμα και δίνοντας κίνητρα για διεπιστημονικές αντιμετωπίσεις. Αυτό μπορεί να μην αρκεί όμως για να επιληφθεί αυτή η δυσκολία την οποία έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις πιθανές επιπτώσεις τις οποίες κάνει ο καθένας στην διεθνή ασφάλεια των τροφίμων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να προωθήσουμε την σωστή γνώση και κατανόηση του σωστήματος των τροφίμων και τον σεβασμό απέναντι στα τρόφιμα μέσω εκπαίδευσης, ε, μέσω επικοινωνίας, έτσι ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν ε, τις επιπτώσεις των προσωπικών τους επιλογών. Κυρίες και κύριοι, το να διατρέφει τον πλανήτη κανείς είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο και περίπλοκο. Πρέπει να το μελετήσουμε σωστά, πρέπει να προβλέψουμε καλύτερα. Εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους έξι μήνες που έχουμε μέχρι το 15 την έκθεση γιατί τότε η προσοχή του κόσμου θα στραφεί προς εμάς έτσι ώστε να κάνουμε προτάσεις απτές και σημαντικές για διεθνή συνεργασία και για καλύτερη ασφάλεια στον τομέα των τροφίμων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσλερ. Καλό θα ήταν να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Χανιώτη από τη Γενική Διεύθυνση για τη Γεωργία να λάβει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Χανιώτη. Thank you, Mr. Chairman. I would be brief. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομό και θα ήθελα να διευκρινίσω αυτή εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην Expo Μιλάνου υπό την πολύ ικανή ε, αιγίδα του σχετική γενική διεύθυνση και διοργανώνουμε πολλές σχετικές εκδηλώσεις. Στην Γενική Διεύθυνση Άγκρη θα έχουμε πάνω από 20 εκδηλώσεις που θα συνδέονται με αυτό και θα ήθελα να επικεντρωθώ εν συντομία σε μία από τις προτεραιότητες τις οποίες ανέφερε και ο κύριος Φίσλερ το θέμα της βιώσιμης διαφοροποίησης η οποία η οποία συνδέεται με τις ε, συζητήσεις που έχει κάνει και η Επιτροπή σας. Ένα από τα θέματα τα οποία θέτουν δύο θέματα αντιφατικά. Βιωσιμότητα και αντιδικοποίηση, η οποία συνεπάγεται και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς και συνέπειες. Μπορεί να διαφωνούμε για το πώς τοποθετούνται, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση προς την χρήση ε, από το κοινό και της ε, γης. Η εντατικοποίηση μας φέρνει στο μυαλό, πιο πολύ τη χρήση των πόρων με τρόπο που μεγεθύνει την απόδοση και την αποδοτικότητα. Το πώς λοιπόν συνενώνουμε τα δύο αυτά στοιχεία με έναν τρόπο συμπληρωματικό, αυτό αποτέλεσε το αντικείμενο πολλών συζητήσεων και στην ε, πρόσφατη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για το μέλλον. Θα πρέπει να οργανώσουμε λοιπόν τουλάχιστον μία εκδήλωση στην έξπο του Μιλάνου που θα επικεντρωθεί σε τέτοια θέματα, να προσπαθήσουμε να βρούμε όχι μόνο την κατεύθυνση που δίνουμε από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου φαίνεται να κινούνται σε παρόμοιες κατευθύνσεις, όπου ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Να υπάρξει σύνδεση με την έρευνα που γίνεται ε, εκτός ακαδημαϊκού κόσμου, αλλά και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες και την δράση του Κοινού Ρευνητικού Κέντρου. Αυτή είναι λοιπόν η γενική κατεύθυνση και συνεργαζόμαστε και με κάποια μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Άρχεται η συζήτηση τώρα. Ο κύριος Δεκάστρο, παρακαλώ γιατί παρακολουθείτε εκ του σύνεγγυς ε, τη διοργάνωση αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Σεκεύσκη, πρόεδρε Σεκεύσκη. Είναι μεγάλη χαρά που βλέπουμε εδώ τον Φραντς Φίσλερ και τον David Wilkinson επίσης. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή την οποία έχουμε μπροστά μας σήμερα ε, και αυτή που μας δίδεται στη χώρα μου, στο Μιλάνο, όχι μόνο για τη χώρα μου αλλά και για την Ευρώπη να μπορέσει να πάρει μέρος στην διεθνή έκθεση γύρω από το θέμα της διατροφικής ασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο όπως και σήμερα το πρωί ε, μας είπε ο Φραντ Φίσλερ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στα πλαίσια της περιγραφής των εργασιών της Διοικητικής Επιτροπής. Το ίδιο συζητάμε και εμείς στην Κομάγκρη τώρα να δούμε ποιες είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες αυτή η Επιστημονική Επιτροπή κατάφερε να συνδυάσει και να εφαρμόσει αυτούς τους πρώτους μήνες εργασίας. Έχει μεγάλη σημασία να αξιολογήσουμε σωστά την προσπάθεια η οποία γίνεται, προσπάθεια εντοπισμού των βασικών στόχων κοινών στόχων και προκλήσεων για το σύνολο του πλανήτη. Ζούμε θα έλεγα στα πλαίσια μιας συγκυρίας που βλέπει τις τιμές των γεωργικών προϊόντων να είναι χαμηλές και ιδιαίτερα μετά από τη συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί για τα, τις τιμές των γαλακτοκομικών κάτι το οποίο γνωρίζει ο κύριος Φίσλερ, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πίεση στις τιμές και μειούνται οι τιμές ε, και προσπαθούμε να δούμε ότι όχι μόνο εμείς αλλά και πως το σύνολο του κόσμου θα μπορέσει να δώσει μια απάντηση σε αυτή την αύξηση της ζήτησης στον τομέα των τροφίμων από την Ινδία, την Ασία μάλλον από την Κίνα αλλάζουν τα καταναλωτικά pattern με ριζικό τρόπο και είναι δύσκολο να δούμε πώς στο μέλλον θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις διατροφικές ανάγκες ε, που ζητά κυρίως ζωοτεχνικά προϊόντα, δηλαδή τεράστιες αυξήσεις στον τομέα καλλιεργιών όπως το αραβόσιτο και η σόγια. Λοιπόν, όπως είπε και ο Φίσλερ, πρέπει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της διατροφικής αλυσίδας, να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και ελπίζω όπως είπε και ο Φίσλερ, ε, στη συνάντηση που θα κάνουμε στο Μιλάνο τον μήνα ε, Ιούλιο του 2015 να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιες πρώτες απαντήσεις σε αυτά τα δύσκολα ερωτηματικά. Εποφελούμε εδώ της παρουσίας του ούτε Επιτρόπου, έτσι ώστε να κάνω μια ερώτηση την οποία ε, μάλιστα επανέφερε ο Τάσος Χανιώτης πριν από μένα. Πώς θα μπορέσει κανείς να αυξήσει τις αποδόσεις και ταυτόχρονα να διαχειριστεί με αηφόρο τρόπο τους φυσικούς πόρους. Μιλήσατε εσείς για αηφόρο εντατικοποίηση. Ακούγεται λίγο αστεία αυτή και να πω λίγο αντιφατική αυτή η ιδέα. Ε, στην ουσία γνωρίζουμε ότι το μέλλον της έρευνας είναι αυτό που θα καθορίσει το συγκεκριμένο πεδίο. Μπορείτε, Πρόεδρε Φίσλερ, να μας δώσετε ε, κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το θέμα αυτό το οποίο θα απασχολήσει πολύ την έρευνα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ράνς Γκαρσία έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά μετά από μία δεκαετία ξαναβλέπουμε τον ε, κύριο Φίσλερ και βλέπω ότι είναι ακμεότατος, όπως το θυμόμαστε όταν ερχόταν στην Επιτροπή μας ως Επίτροπος. Έχω κάποιες ερωτήσεις για την Επιστημονική αυτή Επιτροπή, για την Expo του Μιλάνου του 2015. Μια και πρόκειται για Επιστημονική Επιτροπή που αφορά την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, θα ήθελα να ρωτήσω αν στη συμπερίληψη των θεμάτων της ΕΞΠΟ λάβατε υπόψη το ρόλο των οργανισμών ελέγχου των τροφίμων και ολόκληρη την διατροφική αλυσίδα αν θα ληφθούν και αυτά τα θέματα υπόψη και αν θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Γιατί από τις πιο καινοτόμε εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι ο ρόλος των ελεκτικών οργανισμών και η λήψη υπόψη της διατροφικής αλυσίδας στο σύνολό της, προκειμένου να προστατεύσουμε ε, τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη και την ποσότητα και την ποιότητα ε, των τροφίμων. Ε, πρόσφατα έχουμε θεσπίσει έλεγχο και σχετικές διατάξεις στην Ισπανία για το θέμα αυτό και μετά και το ρωσικό εμπάργο το θέμα γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο. Θα τα λάβει αυτά υπόψη η έξπο του Μιλάνου. Επίσης, ε, θέμα χρηματοδότηση. Από πού θα προέλθουν τα κονδύλια για την έξπο του Μιλάνου, μπορείτε να μα το διευκρινίσετε, γιατί με τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ ένα από τα ζητήματα που μα ικανοποίησαν περισσότερο είναι ότι καταφέραμε για πρώτη φορά ο αγροεπιστηστικός τομέας ε, να ενεργοποιεί τα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Δεν ξέρω ε, πώς χρηματοδοτήσατε εσείς τις εργασίες σας, ή μήπως από τον ορίζοντα 2020. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δόρφ. Κύριε Στορμαντ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φίσλερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της δραστηριότητα της Επιτροπής. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι όντως αληθεύει στο, ότι στο Μιλάνο θα παρουσιάσουμε το ευρωπαϊκό μας μοντέλο, αλλά πρόκειται για μια παγκόσμια έκθεση και το θέμα δεν είναι απαραίτητα μόνο η ευρωπαϊκή γεωργία, όχι το θέμα είναι η γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αν το θέμα είναι πώς ε, θα θρέψουμε τον κόσμο στο μέλλον, βασικό ζήτημα είναι να δούμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλώντας για την βιώσιμα υφόρο αντατικοποίηση. Θα πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι θα πρέπει σχετικά γρήγορα να μιλήσουμε για τεχνολογίες που αναπτύσσονται σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τον τομέα των τροφίμων, αλλά τις ε, απαρνούμαστε στην Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε τέτοιες καινούργιες τεχνολογίες στον τομέα της γεωργίας. Ποια θα είναι λοιπόν η αντιμετώπιση μας στο Μιλάνο, θα συζητήσουμε τέτοια θέματα. Υπάρχει κάτι γνωστό, κάποια γνωστή προσέγγιση. Για να μην σπαζοκεφαλιάζουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Επίσης θα θέλαμε να ξέρουμε με υπό ποια μορφή θα διεξαχθούν οι συζητήσεις αυτές. Θα υπάρχουν δηλαδή σεμινάρια, συνέδρια εδώ στο Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων θα πρέπει να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και να εντάξουμε στην καθημερινή μας εργασία τα αποτελέσματα του Μιλάνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άγνιου. Κύριε Φίσλερ, δεν θα με θυμάστε. Α, με θυμάστε. Α, από τις επισκέψεις στην Εθνική Ένωση Γεωργών του Ηνωμένου Βασιλείου. Όλος παραδόξως ακολουθώ τον ηρμό του προλαλήσαντος. Δεν το φανταζόμουν. Έχουμε δύο ερευνητικά Ινστιτούτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ένα είναι το κέντρο το ερευνητικό του Τζόνανες, είναι και τα δύο στην περιοχή μου και κατάφεραν να βγάλουν πατάτες που αντιστέκονται σε ένα παράσιτο της πατάτας, που είναι μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Πρόκειται για ένα μύκητα που είναι ανθεκτικός στα μυκητοκτόνα και βρήκαν στο Ινστιτούτο αυτό μια λύση χάρη στη γενετική μηχανική. Αλλά ε, ακριβώς επειδή πρόκειται για γενετικό στροπημένο οργανισμό δεν μπορούν να το θέσουν στην αγορά. Και στο Ρόθεμστετ έχουμε άλλο ερευνητικό κέντρο. Εκεί βρήκαν τρόπο να αποτρέψουν το παράστο αυτό από το να σκοτώσει το φυτό. Δεν το σκοτώνει καν δηλαδή το παράστο. Αλλά ούτε και αυτό μπορούμε το το ερευνητικό αποτέλεσμα να το δημοσιεύσουμε γιατί προϋποθέτει και αυτό κάποια γενετική ε, τροποποίηση. Δεν ξέρω αν ε, θα έχουν ένα περίπτερο στο Μιλάνο. Και επίσης ε, μιλήστε για την βιώσιμη την αηφόρο εντατικοποίηση, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύσαμε κάτι πολύ χρήσιμο για τους γεωργούς χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση. Το θέμα της ελεκράμβης, για παράδειγμα, που ε, δυστυχώς δεν μπορούν πια να χρησιμοποιήσουν τους παλιούς πόρους ελαιοκράβης, αλλά νέους φόρους που δεν είναι αρκετά ανθεκτικοί. Οπότε τελικά χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τόσο έντονα εντομοκτώνα που σκοτώνουν το ίδιο το φυτό. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα και στην Βρετανική Γεωργία και στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή αλλά εμείς εθελοτυφλούμε και αποστρέφουμε το βλέμμα από τις λύσεις. Μπορείτε λοιπόν να δώσετε απάντηση σε μένα και στον προλαλήσαντα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Φίσλερ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Η μία για τις ε, αγορές και την αστάθεια των αγορών. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη της ε, γεωργίας είναι επενδύσεις. Και έτσι πως πηγαίνουν αυτή τη στιγμή οι αγορές, υπάρχουν τεράστιες ανασφάλειες και αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά τις τιμές και άρα θα υπάρχει απροθυμία επένδυσης και ήδη διαφαίνεται αυτή η απροθυμία επένδυσης στη γεωργία. Μπορούμε να κάνουμε κάτι στο Μιλάνο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της αστάθειας των τιμών. Κάτι άλλο, το δεύτερο θέμα για τις νέες τεχνολογίες και για την αποδοχή των νέων τεχνολογιών στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αν αποφασίσουμε να μην τις αποτεχτούμε τις νέες τεχνολογίες, τι δυνατότητες έχουμε και επενδύουμε στην έρευνα για να έχουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις, αν αποφασίσουμε ενδεχομένω ότι κάποιες τεχνολογίες δεν μπορούμε να τις αποτεχτούμε. Έχουμε Είχαμε χθε εδώ στο Κοινοβούλιο τον πρόεδρο του IPCC, τον Dr. Πατσάουι. Το μήνυμα προς εμάς ήταν σαφές. Μας είπε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει να παίξει ρόλο η γεωργία, αλλά μιλάει για την εκτενή αναδάσωση των εκτάσεων Άρα, αν αφαιρέσουμε τις εκτάσεις για την αστική ανάπτυξη και για τα δάση, θα έχουμε περιορισμένο χώρο, περιορισμένες εκτάσεις για γεωργία. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή τη βιώσιμη μεταδικοποίηση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι αγορές και οι τιμές θα δράσουν αντίθετα προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα τα δικά σας σχόλια για το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ναι, Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Θα ήθελα και κάποιες απαντήσεις όμως. Γιατί πιστεύω πολύ απλά ότι σε πολλές εκθέσεις έχουμε πάει όπου λέμε ότι όλα είναι καλά και όμορφα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Για παράδειγμα, αν ακούγατε τη συζήτησαμε σήμερα το πρωί για το τομέα της γαλακτοπαραγωγής, θα καταλαβαίνετε ότι τίποτα δεν πάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε τις αντιφάσεις που υπάρχουν για τους ε, συναδέλφους που μίλησαν για τις νέες τεχνολογίες. Εννοείται τη γενετική τεχνολογία. Δεν χρειάζεται παρακαλώ να κάνουμε εδώ πέρα διαφήμιση για αμερικανικού ομίλους. Έχουμε και την ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική και λειτουργεί μια χαρά χωρίς να χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες γενετικές. Η παγκόσμια γεωργική έκθεση και τα άλλα μοντέλα θα πρέπει να παρουσιάσουμε αυτή την αντίφαση που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών πτυχών. Θεωρώ ότι τέτοιες εκθέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες συζήτησης Εδώ και χρόνια συζητάμε στην Ευρώπη για την αντατικοποίηση. Θα πρέπει να συζητάμε και θέματα λοιπόν αντιφατικά. Και όταν μιλάμε για τα τρόφιμα, για το παγκόσμιο πληθυσμό, θα πρέπει να συζητήσουμε και το ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι δεν είναι απαραίτητα οι νέες τεχνολογίες αυτές που θα βοηθήσουν, αλλά χρειάζονται και άλλα μέσα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φεράντι είναι ο τελευταίος μας ομιλητής. Euh, δεν είχα σκοπ... Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, αλλά η παρέμβαση του κυρίου Φίσλερ ε, μου επιτρέπει να συστηθώ κι εγώ, αλλά θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Μας προτείνεται μια φιλοσοφική συζήτηση, θα έλεγα. Ε, το συνδέεται με τον πλανήτη και τις ανάγκες του πλανήτη και προτείνεται τον καλύτερο κόσμο που μπορούμε να έχουμε. Αυτό θα πρέπει να το προτείνεται και στο Παρίσι και στις περιφέρειες γιατί έχουν εξεγερθεί όλες οι περιφέρειες. 5 Νοεμβρίου 100.000 Παραγωγή στην Γαλλία διαδηλώνουν. Διαδηλώνουν γιατί δεν μπορούν πια τις κρίσεις στον τομέα των προϊόντων τους. Μας προτείνεται έναν καλύτερο κόσμο. Αλλά εσείς κύριε Φίσλερ είστε εκτός επαφής με τον γεωργικό κόσμο. Ήσασταν υπεύθυνο για τις διαθετικές πολιτικές και μας κληρονομήσατε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο ε, στην ουσία επιδιώκει την παραγωγή με κάθε κόστος και εκτός ε, των ιδίων των εργαζομένων στη Γεωργία, εκτός των Γεωργών. Ήρθατε εδώ λοιπόν για να ανταλλάξουμε γνώμες και όχι να επιβάλλετε τη δική σας γνώμη. Αλλά εσείς ε, σαν παλαιός επίτροπος πώς μπορείτε να εκπροσωπείτε το μέλλον ε, στο ΕΞΠΟ 2015 εφόσον ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος προώθησε τους στόχους της απορρίθμισης και της απελευθέρωσης. Σπάσατε το γεωργικό μέσο. Πρέπει να πάτε στο Παρίσι να δείτε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική ε, στήρα. Πρέπει να ακούτε το τι πιστεύουν οι βουλευτές που προέρχονται από κράτη τα οποία υποφέρουν από την απορρίθμισή σας. Λυπάμαι για την κατάσταση που μας έχετε αφήσει και εσείς μας προτείνετε το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Ε, όταν σας είχαμε ανάγκη, όταν οι γεωργοί σας είχαν ανάγκη, πού ήσασταν εσείς. Αποτύχατε και τώρα εσείς θα μας δώσετε και συστάσεις για το μέλλον. Και η κυρία pani. το λόγο τελικά. Σας ευχαριστώ κύριε Φίσλερ. Επτά σημεία παρουσιάσατε τα οποία θέλετε να παρουσιάσετε. Τα επτά σημεία σε ό,τι αφορά την, τα τρόφιμα, σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, ποιότητα, όλα αυτά είναι σημαντικά. Μέχρι και την αξιοποίηση των εκτάσεων και την ε, αγροτική παραγωγή, βιώσιμη ανάπτυξη. Στη συζήτηση λοιπόν ακούσαμε πολύ αυτόν τον όρο της βιώσιμης αντιδικοποίησης, της βιώσιμης ανάπτυξης. Αν εστιαστούμε μόνο στην Ευρώπη, θα μείνει μόνο η αντιδικοποίηση. Αυτό κάναμε τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, δυστυχώς το σκέλος της βιωσιμότητας παραμελήθηκε. Αλλά δεν είναι ευρωπαϊκή αυτή η έκθεση, είναι παγκόσμια έκθεση και αν θέλουμε λοιπόν αυτή την βιώσιμη εντατικοποίηση, αν αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε στην έκθεση, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες βιώσιμης εντατικοποίησης και εδώ τονίζω το σκέλος της βιωσιμότητας. Όχι μόνο η οικολογική βιωσιμότητα, αλλά και η κοινωνική βιωσιμότητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η έκθεση για να παρουσιάσει αυτό ακριβώς. Και να μην ξεχάσουμε ότι πρόκειται για μια κερδική έκθεση, γιατί όλα αυτά λοιπόν τα σημεία συμπεριλήφθησαν. Οι ανάγκες έρευνας όλα τα θέματα που αγγίζονται, τα, όλες οι πτυχές του θέματος, θεωρώ ότι είναι σημαντικές. Γι' αυτό, λοιπόν, ήταν τόσο σημαντικό το θέμα της έκθεσης, γιατί όλοι οι σχετικοί φορείς μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Όχι λοιπόν, να μην περιοριστούμε μόνο στην ευρωπαϊκή διάσταση. Είπατε feed the planet όχι we feed the planet, όχι δηλαδή μόνο εμείς στην Ευρώπη να φροντίσουμε για να έχει τρόφιμο ο πλανήτης, για ένα τμήμα μόνο μπορούμε να φροντίσουμε. Και όταν ε, μπορούμε να περάσετε, αν θέλετε, από την ε, επιστηστική ασφάλεια στην επιστηστική επικυριαρχία, θα ήμασταν ακόμα πιο σύμφωνοι μαζί σας. Να κοιτάξουμε τις διάφορες περιφέρειες, λοιπόν, σε μια τέτοια παγκόσμια έκθεση και να μην ε, περιοριστούμε στην ευρωπαϊκή διάσταση, στην ευρωπαϊκή ε, οπτική γωνία. Θεωρώ ότι μόνο έτσι θα ήταν καρποφόρα η εμπειρία και θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και άλλες ιδέες. Πέρα από την ιδέα ότι με οποιαδήποτε καινούργια τεχνολογία μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα της πατάτας ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Οπότε θα παρακαλέσω τον πρόεδρο Φίσλερ να σχολιάσει αυτά που άκουσε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω τώρα στη μετρική μου γλώσσα για να απαντήσω όσο πιο πολλές ερωτήσεις γίνεται, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Μετά θα προσπαθήσω και εγώ λοιπόν να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Να ξεκινήσω από το εξή. Θεωρώ ότι είναι ε, απαραίτητο να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Τόνισα σαφέστατα ότι το έργο της ε, Συντονιστικής Επιτροπής δεν είναι να καταστρώσει μια καινούργια αγροτική πολιτική. Εμείς δεν είμαστε οι πολιτικοί θύνοντες στα πολιτικά όργανα λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι δική σας δουλειά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς αποκλειστικά είμαστε υπεύθυνοι ή αισθανόμαστε υπεύθυνοι αν θέλετε, αφενός κατά την ε, διεθνή έκθεση όλα ή εν πάση περιπτώσει τα πιο πολλά δυνατά σχετικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιστική ασφάλεια να τεθούν και να καταστούν ε, ορατά στην ε, διεθνή έκθεση. Και επίσης, πέραν από αυτό, καθήκον μας είναι ένα, να αναπτυχθεί ένα ερευνητικό το πρόγραμμα, το οποίο θα επικεντρωθεί επειδή δεν είμαστε μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι που εξετάζουμε τέτοια θέματα, αλλά και άλλα τμήματα του κόσμου ρευνούν τέτοια ζητήματα. Να επικεντρωθεί λοιπόν στο ποια θα μπορούσε να είναι η ευρωπαϊκή συμβολή από πλευράς έρευνας, προκειμένου να πετύχουμε το στόχο της επιτιστικής ασφάλειας. Και όλοι ξέρουμε ότι το επόμενο έτος είναι ένα καθοριστικό έτος ως προς αυτό. Γιατί η συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο θα αποφασίσει για το ποιοι θα είναι οι μετέπειτα στόχοι, οι επόμενοι στόχοι μετά τους στόχους της χιλιετίας. Καταρχάς είχαμε θέσει το στόχο της χιλιετίας να μειωθεί κατά το ίμιση ο πληθυσμός που πεινάει. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κατά πάσα πιθανότητα. Ο επόμενος λοιπόν δεύτερος στόχος για τα επόμενα 15 έτη θα είναι να μην υπάρχει καθόλου πείνα. Αυτός ο στόχος είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Και βλέπετε λοιπόν ποιες θα είναι και οι προκλήσεις και για την Ευρώπη. Αλλά στο Μιλάνο μιλάμε για μια διεθνή έκθεση όπου συμμετέχουν 147 χώρες και δεν θα μπορέσουμε να προβλέψουμε και να προδιαγράψουμε για κάθε χώρα το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει. Είναι δική τους επιλογή, είναι απόλυτα ελεύθερες οι χώρες. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κυρίως σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας με την Ιταλική κυβέρνηση που θα έχει και το μεγαλύτερο περίπτερο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει και αυτή δικό της περίπτερο. Τι θέλουμε λοιπόν από κοινού να θέσουμε και να καλύψουμε κατά το δυνατόν όλα τα θέματα που μας αφορούν. Κοιτάξαμε λοιπόν ποιες εκδηλώσεις έχουν διοργανωθεί, έχουν συγγνώμη, προγραμματιστεί ως τώρα. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θεωρούμε ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί προκειμένου ακριβώς να υπάρχει μια συνολική εικόνα. Η συνολική εικόνα την οποία ακούσαμε και την οποία ζήτησαν και διάφοροι βουλευτές άλλωστε. Εν γέννη, ο βασικός, το βασικό σημείο εστίασης είναι το Global Food Security, παγκόσμια επιστηστική ασφάλεια, όπως την ορίζει η ΦΑΟ. Πώς την ορίζει λοιπόν την επιστημιστική ασφάλεια και επιστημιστική ασφάλεια και food safety και θέμα τροφίμων και θέμα ποιότητας τροφίμων. Όλα αυτά αποτελούν σύμφωνα με τον ορισμό της ΦΑΟ μία ενότητα. Κατά δεύτερον, αν θέλουμε αυτό το Global Food Security, αν αυτό είναι ο στόχος, είναι σαφές ότι η παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να αυξηθεί προκειμένου τις επόμενες δεκαετίες να καταφέρουμε να θρέψουμε τα 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η συμβολή κάθε υπήρου και κάθε χώρας δεν είναι η ίδια και απόλυτα σωστά τονίσατε ότι η Ευρώπη εδώ έχει να διδραματίσει πολύ διαφορετικό ρόλο από ότι η Αφρική, η Ασία ή άλλες, σε πάση περιπτώσει, Ήπειροι. Και βάσει των εμπειριών των τελευταίων 70-80 ετών στην Ευρώπη, όπου καταφέραμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάρα πολύ γρήγορα να φτάσουμε σε επίπεδα αυτάρκειας, αλλά τι άλλο μας λέει η ιστορική εμπειρία, ότι αυτή η ανάπτυξη της παραγωγής αφενός προέκυψε από αύξηση και όχι από αύξηση διαθεσιμότητας εκτάσεων. Αυτό τι σημαίνει ότι η αύξηση των ποσών έγινε εις βάρος του περιβάλλοντος σε μεγάλο βαθμό. Όταν τώρα λοιπόν μιλάμε για βιώσιμη εντατικοποίηση, σίγουρα θα υπάρξουν πολλές περιφερειές στην Ευρώπη όπου το θέμα της βιωσιμότητας, άρα δηλαδή της αντιμετώπισης των σφαλμάτων του παρελθόντων, Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί λοιπόν τα ασφάλματα του παρελθόντο και όχι η απαραίτητα μεγαλύτερη παραγωγή. Εκτό αν, ε, αν υπάρχουν μάλλον άλλε περιφέρειε όπου χωρί μεγάλο πρόβλημα και χωρί ιδιαίτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντο μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή, για παράδειγμα σε κράτη τη Αφρική, όπου μπορεί χωρί ε, μεγάλε τεχνολογίε, χωρί ιδιαίτερα προβλήματα, χωρί ε, ιδιαίτερε διαφορέ μπορούν άνετα να διπλασιαστούν οι όγκοι παραγωγής για παράδειγμα στο Μπουρκίνα Φάσο είναι 100 κιλά κατά μέσο όρο η παραγωγή ανά εκτάριο. Άρα το να αυξηθεί αυτό σε 2.000 ε, τόνους, σε 2.000 κιλά, ενώ ο ευρωπαϊκός ε, μέσος όρος είναι 8 τόνοι, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε αυτό το πρόβλημα στην πολυμορφία του, σε όλες τις διαστάσεις, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Και έτσι λοιπόν περνάμε σε διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν. Καταρχάς, το να απαντήσουμε το ερώτημα του πώς μπορούμε βιώσιμα να αυξήσουμε την παραγωγή. Αυτό είναι ένα κλασικό ζήτημα το οποίο είναι διατομεακό. Δεν είναι δυνατόν να το πετύχουμε αυτό μόνο με καλύτερα είδη σπόρων, για παράδειγμα ή ότι λέγοντας ότι πρέπει να αυξήσουμε την απόδοση των ε, γαλακτοφόρων αγελάδων. Όχι, πολλοί παραγόντες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Και ένα από τα σημεία που έχουν να κάνουν με την έρευνα είναι ακριβώς αυτό. Αυτή η ιδιομετωμεακή συνεργασία, δηλαδή η προώθηση τη συνεργασία διαφόρων κλάδων προκειμένου να υπάρξει συνολικά καλύτερη λύση. Σε ό,τι αφορά την κυρία Καρσία, αυτό που ζήτησε, το θέμα των διατροφικών αλυσίδων να παίξει και αυτό το ρόλο του. Αυτό λαμβάνεται υπόψη, σας το λέω ήδη από τώρα, γιατί και εμείς θεωρούμε και εδώ πάλι στην παραγωγική αλυσίδα παίζει το ρόλο της αυτή ότι η συνεργασία των διαφορών τομέων και τα συστήματα των τροφίμων θα πρέπει να μελετηθούν καλύτερα. Όχι μόνο τα μεμονωμένα βήματα της παραγωγής. Όλο το σύστημα λοιπόν. Ο κύριος Ντόρφμαν επέστησε την προσοχή μας στο εξή. Είπε ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και την παγκόσμια διάσταση. Μα ναι, ακριβώς αυτή είναι η πρόθεσή μας. δεν είναι μόνο ενδοευρωπαϊκά τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν. Και γι' αυτό λοιπόν ακριβώς εκείνες τις εκδηλώσεις τις οποίες σχεδιάζουμε στο Μιλάνο και από πλευράς ε, της Συντονιστικής Επιτροπής θα τις προγραμματίσουμε με τέτοιο τρόπο προκειμένου να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την Ευρώπη, γιατί με όλους θέλουμε να συζητήσουμε, με όλους θέλουμε να διεξαγάγουμε διάλογο για το ποια θα είναι η σωστή προσέγγιση σε ό,τι αφορά θέματα έρευνας. Θέλω να πω άμεσα το εξής. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε έρευνα και αυτή την έρευνα να τη θέτουμε υπό τις επιταγές του οποιοδήποτε. Γιατί όταν δεν είναι ελεύθερη η επιστήμη, νομίζω ότι έχει φτάσει στα ωριά της. Η έρευνα και η γνώση δεν σημαίνει ότι δεν έχουν φυσικά κοινωνικό σκοπό και κοινωνικό λειτουργήμα να επιτελέσουν. Όχι βέβαια, αλλά θα πρέπει να επιτρέψουμε στην έρευνα να κινηθεί όπως κινείται. Άλλο θέμα είναι το τι κάνουμε με τα αποτελέσματα της έρευνας. Αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, το οποίο αναπόκειται στην ε, διακριτική ευχαίρεια των πολιτικών αρχών. Αλλά δεν μπορούμε εκ των προτέρων να πούμε και να προδιαγράψουμε ότι επειδή δεν θέλουμε κάτι, απαγορεύουμε την έρευνα στο χύψη τομέα. Αυτό θέτει και μια συζήτηση, νομίζω, και θα έπρεπε να γίνει μια συζήτηση για την δεντολογία την επιστημονική. Και έτσι μπορώ να απαντήσω και σε αυτά που είπε ο συνάδελφος από το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά τις αντιρρήσεις, ε, σε ό,τι αφορά τις διάφορες μεθόδους καταπολέμησης ασθενειών των φυτών. Σε ό,τι αφορά την αστάθεια, την πτυτικότητα, την αστάθεια των τιμών και των αγορών. Αυτό αποτελεί τμήμα της έρευνας και αυτό κυρίως επειδή στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σαφήνεια για το κατά πόσον οι τιμές που ανεβαίνουν ή που πέφτουν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την επιστημική ασφάλεια. Μπορείτε να κοιτάξετε τα σχετικά έγγραφα χαραξής πολιτικής του ΑΣΑ, του ΣΦΑΟ ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Και εκεί θα δείτε ότι πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση το 2008 και 2009, γενικά αυτό που ακούγαμε ήταν ότι για την πείνα στον κόσμο ευθύνονται οι τιμέ που πέφτουν σε όλο τον κόσμο. Το 2010 οι ίδιοι οργανισμοί έρχονται και μας λένε ότι οι τιμές που ανεβαίνουν φταίνε για την πείνα στον κόσμο. Αυτό νομίζω καταδεικνύει πόσο πολύ σύνθετο είναι το πρόβλημα. Πολύ πιο πολύ σύνθετο από ό,τι παρουσιάζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Και αυτή την ε, περιπλοκότητα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε λοιπόν. Αυτό που είπε ο συνάδελφο, ο φίλος μου Πατσάουρη για την ε, αναδάσωση. Τα υπογραμμίζω όλα αυτά. Το γνωρίζω λοιπόν καλά και ξέρω τι σκέφτεται. Το θέμα δεν είναι να αναδασώσουμε τις καλύτερες γεωργικές εκτάσεις. Υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο όπου η αναδάσωση επιδεικνύει πολύ καλά αποτελέσματα. Για παράδειγμα σκεφτείτε τη ζώνη Σαχέλ όπου προχωράει το φαινόμενο της ερημοποίησης. Μόνο με αναδάσωση μπορούμε να ανακόψουμε το φαινόμενο αυτό. Πολύ σημαντική η λειτουργία αυτή. Και υπάρχουν και άλλα τμήματα του κόσμου όπου χωρίς κανένα λόγο διαβρώσαμε τροπικά δάση και άλλους βιότοπους που παρόλα αυτά δεν προέκυψαν γεωργικές εκτάσεις. Και εκεί λοιπόν μπορούμε πολλά να κάνουμε. Η αναδάσωση λοιπόν όντως μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή. Αυτό που δεν θα πετύχουμε, σας το λέω κιόλα. δεν καταφέρουμε όλες τις αντιφάσεις του τομέα της γεωργικής πολιτικής και της γεωργίας να τις ε, λύσουμε. Κάτι άλλο πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Καταρχάς, να αυξήσουμε το επίπεδο της ενημέρωσης και της πληροφόρησης. Και αυτό ισχύει ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά τη χορήγηση σωστών απαντήσεων διάφορων αντιφατικών ζητημάτων. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές οι αντιφάσεις να τεθούν ανοιχτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και χωρίς προδιαγραμμένες ιδέες. Μόνο αν υπάρξει ένα τέτοιο διάλογος και αυτό ζητάμε, γι' αυτό διοργανώνονται στο Μιλάνο μια σειρά εκδηλώσεων όπου θα γίνει στοχευμένη συζήτηση. Μόνο λοιπόν αν γίνει τέτοιο διάλογο, θεωρώ ότι θα προχωρήσουμε. Αυτά που είπε ο συναδέλφο από τη Γαλλία για τη φιλοσοφική συζήτηση ε, δεν ε, εκφράστηκα σωστά, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι έθεσα φιλοσοφικά ζητήματα και φιλοσοφική συζήτηση για το θέμα αυτό. Όχι, πολύ πραγματική, πολύ ρεαλιστική είναι η συζήτηση που διεξαγάγουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Και εγώ είμαι μένω ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής. Αλλά αν θεωρείτε ότι εγώ ως Επίτροπος στα 10 χρόνια όπου είχα την ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μόνο που έκανα ήταν να επιδιώκω την απορρίθμιση, είτε δεν καταλάβατε την πολιτική μου, είτε δεν προσέξατε. Αυτό σας το λέω εντελώς ξεκάθαρα. Έξω από τα δόντια. Κυρίες και κύριοι, αυτοί που θέλουν και ζητούν διατροφική κυριαρχία εδώ έχουν δίκιο. Και αυτό θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την έκθεση, γιατί η Επιτροπή μας είναι συνδεδεμένη και παρακολουθεί στενά αυτά τα θέματα. Επίσης, θυμόμαστε πώς είχε κατάσταση στην ε, γεωργική πολιτική όταν εσείς ήσασταν ε, Επίτροπος Γεωργίας και ο κύριος Μπαρνιά, Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί είναι συναφή τα δύο χαρταφυλάκια. Γιατί θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα υπόψη και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Και τότε λύθησαν πολύ καλές προτάσεις και μέτρα για τους Γεωργούς και την υπαίθρο. Σας ευχαριστούμε. Ένα σύντομο πεντάλεπτο διάλειμμα για να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας για το επόμενο θέμα που είναι ακρόαση για την ε, πολιτική των δασών. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσλερ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, περνάμε στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασής μας. Και με μεγάλη χαρά κηρύσω την έναρξη της ακρόασής μας με θέμα την στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργανώνουμε την ακρόαση αυτή για να προετοιμάσουμε την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας που θα καταρτήσει η κυρία Κέστιγκερ. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για τη νέα δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2013. Δεν καταφέραμε όμω τότε να επιληφθούμε δεόντως του θέματος αυτού εξαιτίας ε, των επικείμενων ευρωεκλογών τότε. Εξού και η καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τη νέα στρατηγική για τα δάση. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Ολοκληρώσαμε, διοργανώσαμε λοιπόν αυτή την ακρόαση θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Κέστιγκερ που είναι η συγγήτριά μας. Επαναλαμβάνω θέμα, είναι η νέα στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα στην κυρία Κέστιγκερ για να μας κάνει την εισαγωγή και κατόπιν θα ακούσουμε τις παρουσιάσεις των καλεσμένων μας, τους οποίους και καλωσορίζω εγκάρδια. Θα τους δώσω σε λίγο το λόγο για να μας παρουσιάσουν τα θέματά τους. Κυρία Κέστιγκερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σύντομη γιατί το σημερινό απόγευμα είναι αφιερωμένο και θα έπρεπε να είναι αφιερωμένο στους εμπρεογνώμονές μας, τους οποίους και ευχαριστώ που ήρθαν σήμερα στην Επιτροπή μας για να μας μιλήσουν για το τόσο σημαντικό θέμα της δασικής στρατηγικής μαζί με εμάς, με τους ευρωβουλευτές. Είναι, θεωρώ, ένα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τέλη Σεπτεμβρίου έγινε μία δήλωση με της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το νέο εκλεχθέν Ευρωκοινοβούλιο και είμαστε κάπως καθυστερημένοι. Το Συμβούλιο έχει τοποθετηθεί ήδη για τη στρατηγική αυτή. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να δώσουμε πληροφόρηση ευρεία στους βουλευτές σε ό,τι αφορά την πρακτική πλευρά της πολιτικής αλλά και την επιστημονική πτυχή. Και νομίζω την τελευταία εβδομάδα κατέστησα σαφές με το ενδιαφέρον που εκφράστηκε ποια είναι η σημασία του δασικού τομέα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα δάση αποτελεί και μια πηγή απασχόλησης, ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, είναι μεγάλη η συμβολή του και σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα αριθμητικά στοιχεία μιλούν από μόνο τους. Ως Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να υπερψηφίσουμε μια φιλόδοξη στρατηγική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την εμπειρογνωμοσύνη σας και αν να ακούσουμε τα σχόλιά σας και τις εισηγήσεις σας. Μετά αυτή τη σύντομη παρουσίαση περνάμε στο πρώτο τμήμα της ακρόασης για την πολιτική των δασών και τις θέσεις απασχόλησης. Πρώτος θα λάβει το λόγο ο κύριος Χάραλτ Μάουζερ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών και κατόπιν ο κύριος Χακαράινεν από το Φιλανδικό και η Κεντρική Ένωση Γεωργικών Παραγωγών και Ιδιοκτητών Δασικών Εκτάσεων. Παρακαλώ κύριε Μάουζερ, έχετε το λόγο. Θα στήμασταν ευγνώμονες αν δεν ξεπερνούσατε το χρόνο σας. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like... Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω σαν Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την συγκεκριμένη ακρόαση. Η στρατηγική για τα δάση του 2020 και οι στόχοι για τα δάση του 2020 είναι η βασική συνεισφορά των δασών στην οικονομία γενικότερα. Τα δεδομένα τα οποία σας παρουσιάζω παρουσιάζουν ε, κάποια στοιχεία οικονομικά για τον τομέα αυτό τα οποία η τελευταία τους ενημέρωση και είναι πλήρως ενημερωμένα ε, μέχρι το τέλος του 2011. Βέβαια έχουμε ελλείψεις για τον αριθμό των ιδιοκτητών, των 11 εκατομμυρίων ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, τα θέματα της χρήσης για την παραγωγή ενέργεια, για τα βιοχημικά, τα ε, βιοϊφάσματα είναι πράγματα τα οποία ελείπουν από τις στατιστικές γιατί δεν θεωρείται μερικές φορές ότι ανήκουν στις στατιστικές του δασικού τομέα. Παρ' όλα αυτά μπορεί κανείς λοιπόν να πει ότι τα στατιστικά δεδομένα υποτιμούν εν πολλής και μάλιστα σε ορισμένους τομείς σοβαρά ε, το πραγματικό μέγεθος. Πιστεύουμε λοιπόν ότι στα πλαίσια της νέας στρατηγικής θα καλυφθούν τα κενά αυτά από τα διαθέσιμα στοιχεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουν το τμήμα της βιομηχανίας το οποίο μας δείχνει το σχετικό μέγεθος του τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια σύγκριση ανάμεσα στις πέντε μεγαλύτερες βιομηχανίες. Ε, η δασική βιομηχανία έχει τις ε, περισσότερες εταιρείες, το 1 τρίτο των θέσεων απασχόλησης, και προσφέρει προστιθέμενη αξία περισσότερη από τη χημική βιομηχανία και λίγο λιγότερη από την αυτοκινητοβιομηχανία. είναι θα έλεγα ε, είμαστε εμείς ο βασικός χώρος, ο πράσινος βασικός χώρος της οικονομίας και της βιομηχανίας. Η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτήν την σημασία με συγκεκριμένα μέσα προσανατολισμού. Είναι ένα από τα έγγραφα τα οποία σας έχουμε καταφέσει. Ποιος κανονικά τώρα καλείται να ωφεληθεί από τον συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν τομείς όπως ε, η ε, συλλογή του ξύλου, ε, οι ίδιοι ιδιοκτήτες, η επεξεργασία των προϊόντων ξύλου και άλλα τμήματα της βιομηχανίας που παρέχουν αρκετές δυνατότητες. Αλλά για τον υπόλοιπο τομέα ε, βρίσκονται όχι τόσο σε περιοχές υπαίθρου αλλά σε αστικές περιοχές, δηλαδή βιοενέργεια, οικοσυστήματα, Γενικά σε πάρα πολλούς τομείς οι υπηρεσίες γύρω από την δασική παραγωγή προσφέρονται σε αστικές περιοχές περισσότερο παρά σε περιοχές της υπαίθρου. Ο τομέας αυτός ο δασικός λοιπόν δίνει δυνατότητες ανάπτυξης και για τις αστικές περιοχές και για τις περιοχές της υπαίθρου. Δεν έχουμε όμως όπως είπα τα σωστά στατιστικά στοιχεία για το αστικό κομμάτι έχει ενδιαφέρον να δούμε τα στοιχεία αυτά, ιδιαίτερα για το μέλλον. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη μορφή συντονισμού και για άλλες πολιτικές πέραν της πολιτικής ε, γεωργίας, στον τομέα της γεωργίας. Αυτά τα οποία είπα μέχρι τώρα αφορούν περισσότερο το παρελθόν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τρέχουσες αλλαγές. Ο τομέας, ο δασικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην φάση που θα χαρακτήριζα της δημιουργικής καταστροφής. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες από τις οικονομικές δραστηριότητες μειούνται, ενώ ταυτόχρονα νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες όπως και νέα επιχειρηματικά πρότυπα αναδύονται. Αποτέλεσμα είναι ότι, ε, έχει, ε, θα αλλάξει, ότι θα αλλάξει ο τομέας στις επόμενες δύο δεκαετίες παρά τον προηγούμενο αιώνα. Θα υπάρξουν ε, πολύ περισσότερα προϊόντα, μεγαλύτερη ενεργειακή ε, αποδοτικότητα ε, και οι υπηρεσίες θα συνδέονται καλύτερα με τους υπόλοιπους τομείς. Πολλές από τις αλλαγές αυτές θα έλεγα δεν τις βλέπουμε στις παρούσες έρευνες και στα στοιχεία. Η στρατηγική, η δασική μπορεί να βοηθήσει τον τομέα έτσι ώστε να βοηθήσει την ευημερία των παραγωγών και των γεωργών στην Ευρώπη, αλλά αυτό προαπαιτεί θα έλεγα την σωστή κατανόηση των αλλαγών που επέρχονται. Η βιομηχανία αυτή συνδέεται άμεσα και με τις υπόλοιπες πρώτες ύλες και την επεξεργασία των πρώτων υλών και αποβλήτων. Η αλληλοσύνδεση αυτή εξαρτάται από την προμήθεια θα έλεγα πρώτων υλών από τα δάση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά των δασών, αλλά όλα τα δάση αυτά μπορούν να παρέχουν μέσα και να προκαλέσουν συνέργειες ανάμεσα στις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρουν. Και κάποιες επίσης ε, αλλαγές και περιορισμοί μπορεί να υπάρξουν σε σχέση ε, με τον περιορισμό των ποσοτήτων τα οποία, οι οποίες μπορεί να υλοτομηθούν σε αιτήσια βάση. Αλλά παρόλα αυτά τέτοιες ε, περιοριστικές τάσεις πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά γιατί μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση. Έχουμε ένα παράδειγμα στην περίπτωση της Αυστρίας το 10% στην παρούσα φάση είναι ε, τομέας και χώρος μη παρέμβασης. Αυτό οδήγησε ε, σε απώλεια θέσεων απασχόλησης που εκτιμάται από 6 μέχρι 31% του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού. Αυτό είναι ένα επιχείρημα όχι υπέρ κατά της νέας μορφής διαχείρισης αλλά υπογραμμίζουν την μεγάλη σύνδεση ανάμεσα στο πλαίσιο διαχείρισης και την ίδια τη βιομηχανία και καλείται εδώ θα έλεγε ο καθένας να δει ακριβώς πώς συνδέεται γενικότερα η περιφερειακή οικονομία με τον δασικό τομέα. Στο μέλλον θα υπάρξουν και νέα προϊόντα και υποπροϊόντα από το δάσος που παρέχουν νέες δυνατότητες ε, χρήσιμες για την οικονομία και για την επίτευξη των πολιτικών μας στόχων όπως ε, η απασχόληση, η δημιουργία θέσεων εργασίας δηλαδή και άλλα. Απαιτούνται πολιτικές βέβαια σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διευκολύνουν τις νέες αυτές χρήσεις και τις νέες παραγωγές η βιοπικιλότητα, η πολιτική στον τομέα της μετρίασης των κλιματολογικών αλλαγών και η αηφορία είναι χαρακτηριστικά απαραίτητα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μας οδηγήσουν να αγνοήσουμε το τεράστιο δυναμικό του δασικού τομέα μιας ε, οικονομικής δραστηριότητας με χαμηλή παραγωγή ε, αδιοξιδίου του άνθρακα. Κάποια συμπεράσματα τώρα. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε ότι όταν λαμβάνουμε μία απόφαση για ένα τμήμα του τομέα να βλέπουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στον υπόλοιπο τομέα και όχι μόνο για τα δασικά, δεν αναφέρομαι αποκλειστικά εδώ στον δασικό τομέα γιατί επηρεάζεται γενικότερα η οικονομία ε, της υπαίθρου. Για να το κάνουμε αυτό απαιτείται να έχουμε καλύτερη γνώση των συστημάτων των δασικών Πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στα δάση μέχρι τώρα και να βλέπουμε επίσης και κάποιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των συστημάτων διαχείρισης. Δεύτερον, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν σαν κίνητρα έλξης για επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ο τομέας το δασικός θα πρέπει να είναι πιο ελκυστικός και για τους νέους σε ηλικία ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, σε επιχειρηματίες ε, οι οποίοι ε, θα φέρουν με τη σειρά τους επενδυτές που τόσο χρειάζεται ο τομέας για να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να καταστεί μια βιώσιμη οικονομία. Τρίτον, η έρευνα και η καινοτομία σε κάθε επίπεδο είναι κάτι το κρίσιμο για το σύνολο του τομέα και κυρίω για αυτούς οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν. Απαιτείται ο συνδυασμός των επιστημονικών τομέων, απαιτείται έρευνα πιο στοχευμένη που να οδηγεί σε καινοτομικές μεθόδους εκμετάλλευσης, λόγω της περιπλοκότητας του τομέα και λόγω της τεράστιας γκάμας διαφορετικών δραστηριοτήτων οι ερευνητικές δραστηριότητες είναι πολύ διασπασμένες και μοιράζονται σε πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ένας, ένα πρόγραμμα Horizon 2020 στοχευμένο για την δασική δραστηριότητα να πω ότι στις 13 Νοεμβρίου του 2014 θα οργανωθεί εδώ στο Κοινοβούλιο μια εκδήλωση για τα μελλοντικά βήματα στα δάση και την λεγόμενη βιοοικονομία. Έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε περισσότερα για τις επερχόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στις δασικές περιοχές. Σας ευχαριστούμε. prelegenta. Bardzo Θα δώσουμε τώρα το λόγο στο δεύτερο καλεσμένο μας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, σας ευχαριστώ για την ε, λαμπρή ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δάση, τον κλάδο και τις θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα πρώτα να επισημάνω ότι οι διοκτήτες δασικών εκτάσεων στη Φιλανδία αλλά και στην Ευρώπη γενικώ ε, χαιρετίζουν θερμά την νέα στρατηγική και είμαστε ιδιαίτερος ευγνώμονες για την ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους στα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι όταν μιλούμε για τους κλάδους αυτούς, του συναφείς με τη δασοκομεία και τις θέσεις απασχόλησης, στη Φιλανδία και στην Ευρώπη έχουμε πραγματικά τεράστια αποθέματα βιώσιμων ε, φυσικών πόρων που αυξάνονται συνεχώς. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία η αύξηση του ξυλαποθέματος Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ακριβώς όπως το σύνολο της Φιλανδίας. Μόνο 60% της ετήσιας αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται σε εκμετάλλευση. Και ήταν σχετικά σταθερή κατανάλωση στρογγυλής ξυλίας. Οπότε η βιώσιμη εκμετάλλευση μπορεί να αυξηθεί κατά 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Πόρους έχουμε και μάλιστα α, βιώσιμους πόρους, αϊφόρους. Θα ήθελα να επισημάνω ε, τις χθεσινές ε, προβλέψεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προπτική ανάπτυξη του κλάδου ε, του οικονομικού κλάδου, που είναι μεγάλη πρόκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι οικονομική ανάπτυξη, οικονομική ευμάρεια. Όπως και η επιστολή ανάθεση καθηκόντων του κυρίου Γιούνκερ προς τον Επίτροπο Γεωργίας, ε, πιστεύουμε ότι το επίκεντρο ε, των προσπαθειών για το μέλλον της ε, γεωργίας και της ανάπτυξης υπαίθρου θα πρέπει να είναι η δημιουργία επενδύσεων και θέσεων απασχόλησης προκειμένου να δημιουργηθεί οικονομική ανάπτυξη. Και από αυτήν την άποψη ο δασικός κλάδος θα διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον της βιοοικονομίας. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικό και ισχυρό δασικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσελκύει επενδύσεις και καινοτομία για να μπορέσει να πραγματώσει αυτή την οικονομική ευμάρεια που δεν θα γίνει μία νυχτή ούτε ως διαμαγεία. Το μείζον ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχουμε πολλές πολιτικές ε, που σχετίζονται με την ε, δασοκομεία. Κλιματικές αλλαγές, ε, βιοπικιλότητα, ενέργεια και οι πολιτικές αυτές επηρεάζουν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στη δασοκομεία. Τώρα με την έυτη στρατηγική για έχουμε πολύ καλό σημείο αφετηρίας για να βελτιώσουμε την συντονιστική των πολιτικών που αφορούν τα δάση και να βελτιώσουμε και τον συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε βιοπικιλότητα, πράσινες υποδομές, την Σύμβαση για τη Βιολογική Βιοπικιλότητα, παράνομη υλοτομία, την οδηγία για τα διαιτήματα τα πτηνά. Έχουμε πια πολύ καλούς μηχανισμούς και μέσα για να βελτιώσουμε το συντονισμό των επιμέρους πολιτικών. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, η νέα στρατηγική για τα δάση μπορεί να προσφέρει απτά μέσα για τη μελλοντική μας ευημερία. Όπως είπε πριν από λίγο ο κύριος Μάζερ, σήμερα η δασοκομεία και οι συναφείς κλάδοι απασχολούν 4 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους, κυρίως στις αγροτικές ζώνες και παράγουν ξύλα, ξυλία και άλλα αγαθά με συνολική αξία 500 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 8% του ευρωπαϊκού μεταποιητικού ΑΕΠ και έχουμε εκατομμύρια ιδιωτών δασικών ιδιωτικών δασών που παράγουν ξυλία και συμβάλλουν σε αυτή την ευημερία. Από την άποψη των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, ο ρόλος των ανανεώσιμων φυσικών πόρων και οι λύσεις θα πρέπει ε, που στηρίζονται σε αυτές θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά στο μέλλον και η αύξηση της χρήσης του ξύλου και της ξυλίας θα έχει πολύ θετικές και πολύπλευρες συνέπειες και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι συναφείς με τη δασοκομεία κλάδη θα πρέπει να χρησιμοποιούν κυρίως ε, τοπικά υλικά και έτσι θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από εισαγόμενες πρώτες ύλες. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο της παραγωγής γιατί η παραγωγή αυτή χρησιμοποιεί κυρίως εγχώρια υλικά και εγχώριες πρώτες ύλες. Παρ' όλα αυτά, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτούς τους φυσικούς πόρους, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τα δάση μας και την ξυλία μας, για να εξασφαλίσουμε στο μέλλον οικονομική ευμάρεια θα πρέπει να δείξουμε πολιτική βούληση και ανοιχτό μυαλό. Οι πολιτικοί θύνοντες ε, θα πρέπει να δείξουν αυτή τη βούληση και το ανοιχτό μυαλό. Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δάση. Δεν θα έχει εφαρμογή. Αν δεν έχει, ε, δεν έχει αυτή η εφαρμογή θα είναι απλώς ε, ωραία λόγια και ευχολόγια θα πρέπει η στρατηγική να συμβάλλει στην ε, δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης. Και γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή. Αυτή είναι το κλειδί. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε μέτρα και δράσεις που θα συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης ε, και στην ε, εξασφάλιση της ευημερίας στην Ήπεθρο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει το πολιτές σχέδιο εφαρμογής που θα έχει θεμελιώδη σημασία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πολιτές εφαρμοστικό σχέδιο να περιλαμβάνει χειροπιαστά μέτρα και μηχανισμούς για να μπορέσουμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε τα δάση μας για να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη και οικονομική ευημερία. και να δημιουργήσουμε μια βιοοικονομία στην Ευρώπη που θα στηρίζεται στη δασοκομεία. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε οι πολιτικές και οι νομοθεσίες να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ε, να μην προσθέτουν ε, επιπλέον κόστος και γραφειοκρατία στον κλάδο. Και όταν μιλάμε για την νέα για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θέσεις απασχόλησης, και τις οικονομικές πτυχές και τους συναφείς κλάδους, θα πρέπει να διαρωτηθούμε. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ρυθμίσουμε τις διαφορετικές χρήσεις του ξύλου. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε περισσότερη ρύθμιση για τη βιοπικιλότητα. Γιατί η βιοπικιλότητα, οι κλιματικές αλλαγές, ο ρόλος των δασών στις κλιματικές αλλαγές είναι πολύ σημαντικά θέματα κέρια σημασία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν και αυτές τις αξίες. Όταν όμως μιλούμε για τους κλάδους και τις α, θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να διαρρευθούμε αν χρειαζόμαστε περισσότερες διατάξεις για την βιοπικιλότητα. Χρειαζόμαστε κριτήρια υφόρου διαχείριση δασών για την ευρωπαϊκή παραγωγή αν δεν μπορούμε να πετήσουμε παρόμοιους κανόνες από τις τρίτες χώρες. Κατά τη γνώμη μου, και κατά τη γνώμη των ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να διευρύνει το ρόλο των δασικών κλάδων και τη συμβολή τους στην ευρωπαϊκή οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Το θέμα είναι πώς θα προωθήσουμε τη χρήση του ξύλου και της ξυλίας. Γιατί με το ξύλο μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα αυτά που κάνουμε χρησιμοποιώντας το πετρέλαιο. Χρειαζόμαστε ένα νέο καινοτόμο τρόπο σκέψης, πιο ευρηματικό και δημιουργικό, προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτή τη νέα οικονομία στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Po, tych dwóch Ακούσαμε τους δύο πρώτους καλεσμένους μας και θα έχουμε τώρα ένα γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο της ακρόασης. Παρακαλώ λοιπόν, τι αγορεύει βούλετε. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις ε, στους καλεσμένους μας για το πρώτο τμήμα της ακρόσης που αφορά την δασοκομεία και τις θέσεις απασχόλησης. Πρώτη ζήτηση το λόγο η συγκεκριά μας, η κυρία Κέστιγκερ. Παρακαλώ και περιμένω και τους υπόλοιπους συναδέλφους όσους θέλουν να λάβουν το λόγο και να θέσουν ερωτήσεις να το δηλώσουν. Μην ξεχνάτε ότι θα έχουμε και δεύτερο γύρο ακρόασης και θα έχουμε την ευκαιρία και στο δεύτερο γύρο να θέσουμε ερωτήσεις και να λάβουμε απαντήσεις. Παρακαλώ κυρία Κέστιγκερ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι ο κύριος Μάζερ μίλησε για το δασικό τομέα και είπε ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι ελκυστικό και για τους νέους δασοκόμους. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω κατά πόσον υπάρχουν ε, πρωτοβουλίε στα διάφορα κράτη-μέλη, κυρίως για τη νέα γενιά, προκειμένου να υπάρξουν κίνητρα Ξέρω για παράδειγμα από πλευρά της Αυστρία ότι υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση σε ό,τι αφορά τη διαβίου κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Και θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις θέσεις εργασίας, κατά πόσον υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία, κατά πόσον το δυναμικό ανάπτυξη αυτών των πράσινων θέσεων απασχόληση είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί αριθμητικά. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και θα θέλαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προ την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερως σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία στην Ήπεθρο. Γιατί όλε οι περιοχέ που είναι μακριά από τα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν από την αστιφιλία και εδώ πέρα θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να, να προσφέρουμε λύσεις. Σας ευχαριστώ. Κύριος Έριξον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που αναφέρθηκαν. Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο αυτό που πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ωστόσο, κάποια πράγματα θα μπορούσαμε να τα εξετάσουμε πιο πολύ εις βάθος. Ένα συναλλικό ερώτημα. Είναι το εξής. Εξετάζοντας τον δασικό κλάδο στην Ευρώπη και την σχετική οικονομία, αλλάζει ο κλάδος αυτός. Υπάρχουν ε, νέα υφάσματα. Το χαρτί μειώνεται αποτελεί μικρότερο κομμάτι της συνολικής οικονομίας. Η ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ξύλο των δασών για πολλούς και διαφορετικούς σκοπούς στο μέλλον. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κάποια βεβαιότητα σε ό,τι αφορά το στόχο, το σκοπό όλων αυτών των ερωτημάτων σε εμά τις σκανδιναβικές ε, χώρες, στο βόρειο τμήμα της Ευρώπης, το δάσος αποτελεί μεγάλο τμήμα της ε, χώρας. Σε άλλα τμήματα της Ευρώπης είναι μεγάλη η αποδάσωση. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, νομίζω ότι πριν από 2.000 χρόνια χάθηκε μεγάλο τμήμα των δασών. Αλλά όταν λέτε ότι είστε τόσο θετικοί προς τον δασικό κλάδο, και ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει πιο πολύ μεγάλη δασική έκταση στο μέλλον για πιο πολλές θέσεις απασχόλησης Πιστεύετε λοιπόν, ε, κύριε Μάουζερ και κύριε Χακάνιν, ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό των δασών στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σουλαζό. Ξέρετε, τα ευρωπαϊκά δάση και κυρίως τα γαλλικά αιμορραγούν. Πρέπει να ληφθούν λοιπόν μέτρα άμεσα για να τεθεί Η Κίνα, όπως ξέρετε, διπλασίασε μέσα σε ελάχιστο ε, χρόνο τις εισαγωγές της. Ε, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταναλώθηκαν τεράστιες ποσότητες και δεν έχουμε και πάρα πολλά στοιχεία γιατί ένα μεγάλο τμήμα των προϊόντων αυτών επανεξάγεται στην Ευρώπη υπό τη μορφή παρκέ. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και απειλεί ε, πάρα πολλές θέσεις απασχόλησης σε περιοχές της Γαλλίας όπως το Ερώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη οικονομική δύναμη στον κόσμο που δεν έχει πάρει μέτρα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο το οποίο πλέον έχει έρθει για να παραμείνει. Η Ρωσία, ο Καναδάς, ακόμα και αφρικανικές χώρες έχουν μειώσει δραστικά την εξαγωγή του τρίματος. Ε, μήπως θα πρέπει και εμείς να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ευχαριστώ κύριε Κούσμιουκ. Ο κύριος Μάουσερ στην παρουσίασή του είπε ότι η ξυλία και η δασοκομεία έχει την ίδια σημασία με την αυτοκινητοβιομηχανία. Τι εννοεί ότι έχει την ίδια αξία. Αναφέρεται στον τζίρο, στην αξία του προϊόντος ή έχει κατά νου άλλα στοιχεία μπορείτε να μας αναλύσετε ακριβώς τι εννοείτε όταν λέτε ότι η εντασοκομεία είναι εξίσου σημαντική με την αυτοκινητομηχανία οικονομικά. Ο κύριος Ροπέ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά άκουσα ότι έγινε μια προσπάθεια για να φτάσουμε σε μια συμβαστική λύση και είναι πολύ καλά το παράδειγμα αυτό μιας και ο συμβιβασμός σημαίνει ότι υπάρχουν καλές προπτικές για να καταλήξουμε σε μία λύση. Η στρατηγική εστιάζεται στην δασική ανάπτυξη. Παρά όλα αυτά πρέπει να τονίσουμε ότι στη Λιθουανία η βιώσιμη δασοκομεία θα μπορούσε να προωθηθεί μόνο εφόσον οι συνεταιρισμοί και τα συνδικάτα συμφωνήσουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το καθήκον να ανατεθεί σε επαγγελματίε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αν χορηγηθεί αρρωγή στον κλάδο της δασοκομείας θα πρέπει αυτή η αρρωγή να χορηγηθεί σε συνδικάτα και ενώσεις. Θα πρέπει επίσης να προωθήσουμε συγκεκριμένα ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων της δασοκομείας και πλέον έχει φτάσει θεωρώ η στιγμή να γίνουν συζητήσεις προκειμένου να υπάρξει ανάλογη μεταρρύθμιση στο δασικό κλάδο όπως τον γεωργικό κλάδο. Βλέπουμε σαφή δια... διάκριση εξουσιών και λειτουργιών στον δασικό κλάδο μιας και είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει και η κοινωνική και η οικονομική πτύχη του δάσους. Στη Λιθουανία όμως βλέπουμε ότι όλο και μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στο κλάδο και αυτό σημαίνει ότι συρρυκνώνεται όλος ο κλάδος. Σα ευχαριστώ. κυρία Μοσλιτάιερ. Μακτάιερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσες οι δύο παρουσιάσεις αυτές. να συζητήσω ήθελα τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών ρυθμίσεων στην, στον κλάδο της δασοκομείας. Αν κάτι έχω μάθει τους τελευταίους μήνες ε, που είμαι στις επιτροπές αυτές είναι πως υπάρχουν πάντα παράπλευρες συνέπειες. Πάντα οι προθέσεις είναι οι καλύτερες, αλλά στην εφαρμογή φαίνεται ότι συχνά το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από το ευκταίο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές και να δίνουμε κίνητρα βιωσιμότητας, αλλά όχι πάντα να γίνεται ρύθμιση και ενοποίηση. Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο παράδειγμα επιτρέψτε μου. Η οδηγία για τους βιοτόπους. Στον Εμένα Βασίλειο, η διαχείριση ξυλίας και εκτάσεων που παράγουν ξυλία ε, παρεμποδίζεται από τη σχετική νομοθεσία για τα σβιωτόπους και τελικά ο κόσμος δεν ε, προτίθεται να διαχειριστεί τέτοιες εκτάσεις ε, ξυλίας γιατί φοβάται. Ενώ αν ήταν σωστή η διαχείριση των εκτάσεων αυτών θα ήταν υποφελές αυτό και για τα ενδεμικά είδη. Αυτό φαντάζομαι ισχύει και για άλλες νομοθεσίες. Πείτε μου Λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας για όλες αυτές τις περιβαλλοντικές ε, διατάξεις. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τεράστιο αυτό το θέμα και η δοσοκομεία είναι σημαντικό με της ε, Σουηδική οικονομίας, ε, απασχολεί μεγάλο αριθμό εργαζομένων και είναι σημαντικό θέμα η κοινή στρατηγική για τα δάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά ζητήματα είναι κρεμή. Ε, έχουμε την προστασία φαινός και την παραγωγή φετερού. Είναι αντιφατικές μεταξύ τους έννοιες ή μπορούμε να τις ε, αξιοποιήσουμε και να τις αλληλοσυμπληρώσουμε. Έχουμε και το θέμα της βιοπικιλότητας στα δάση μας. Και Συνεχίζοντα την ερώτηση τη κύρια Μακιντάιερ, ρωτώ, είναι δυνατόν να έχουμε σωστή διαχείριση, με σωστή διαχείριση δασών μεγαλύτερη βιοπικιλότητα από ό,τι αν τα δάση να αναπτύσσονται μόνα τους. Έχουμε πραγματικά ε, μεγάλο αναξιοποιητό δυναμικό των ε, δασών. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα, τα ορυκτά καύσιμα μερικές φορές με τη ξυλία ή να περιορίσουμε ε, τη χρήση του το ε, και σίγουρα έχει, έχουμε αφήσει ακόμη αναξιοποιεί το τεράστιο δυναμικό των δασών γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές ε, εφαρμογές. Και θα υπάρχουν φυσικά μεγάλες διαφορές ε, στη διαχείριση των δασών μεταξύ βορρά και νότου. Έχουμε πολλά ζητήματα λοιπόν να εξετάσουμε και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τη διατύπωση, γιατί όταν μιλούμε για αποψήλωση δασών, σε μερικές χώρες μπορεί να σημαίνει καταστροφή δασών, η υλοτομία. Αλλά στην Σουηδία έχουμε πολύ περισσότερα δάση από μία, πριν από μία πεντηκονταετία, ακριβώ εξαιτία των καλών σχεδίων διαχείριση που εφαρμόζουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε στους κοινούς κανόνες διαχείρισης ίσως ε, με την υπερβολική ρύθμιση κεντρικό επίπεδο αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Γιατί και τα δάση έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των διαφορών χωρών διαφέρουν. Οπότε, καλό θα ήταν η Επιτροπή μας αν ασχοληθεί με την δασική στρατηγική να μπορέσουμε να ε, αυξήσουμε την παραγωγή, την ε, οικονομική ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης. Αν έτσι ε, εξετάσουμε τη δασική στρατηγική, τότε μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τους οικονομικούς αλλά και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Αλλά μερικές φορές έχουμε αποκλίνουσες απόψεις ανάλογα από τη χώρα καταγωγής μας ή από τη ποια πλευρά λαμβάνουμε στη συζήτηση. Και πώς χρησιμοποιούν τα δάση, μόνο για αναψυχή ή για αναψυχή αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παρουσιάσεις αυτές, αλλά πρέπει να πω ότι γενικά υπάρχει αυτή η διάσταση και η εστίαση στην Βόρεια Ευρώπη. Μιλάμε για μια ευρωπαϊκή δασική στρατηγική και να δούμε ότι είναι διαφορετικές οι στρατηγικές για τον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι για το Βορρά ή ακόμα και για τη Γερμανία. Αν δεν απαντήσατε λοιπόν, ίσως θα υπάρχουν άλλες σχετικές παρεμβάσεις και παρουσιάσεις ή μήπως πρέπει να χωρίσουμε σε Βορρά και Νότο την δασική πολιτική. Γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Η μηπω πρεπει να χωρισουμε σε βορρα Μακεντάρ είπε ότι ρώτησε κατά πόσον οι περιβαλλοντικές διατάξεις παρεμποδίζουν την δασική ανάπτυξη. Πρέπει να απαντήσω αρνητικά. Υπάρχουν πάρα πολλέ πτυχέ που πρέπει να λάβουμε υπόψη και η στρατηγική για τη βιοπικιλότητα τη Ευρώπη. Αν μα ενδιαφέρει στα σοβαρά, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτό το 5% από την εντατική καλλιέργεια και αξιοποίηση για βιοτόπους. Θα πρέπει λοιπόν να επιλύσουμε τα θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν που προκάλυψε έκπληξη αυτό που είπε ο κύριος Χάρκαν, ότι δεν θα πρέπει να ενοχικλεί η πολιτική. Νομίζω και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα επί, του, επί της αρχής. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν προβλήματα υπερβολικής ε, αξιοποίησης Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να λεφθούν υπόψη. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την οικονομική διάσταση. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος απάντηση το να αφαιρεθούν όλες οι υπόλοιπες πτυχές και διαστάσεις. Στην βασική στρατηγική Ακούσαμε διάφορα για τις θέσεις απασχόλησης, για τη βιομηχανία, τον οικονομικό κλάδο, αλλά δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο από δική σας πλευρά κατά πόσον πιστεύετε ότι η δασική στρατηγική εδώ ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε και οι δύο πού πιστεύετε ότι είναι τα κρίσιμα σημεία, τα επικριτικά σημεία σε ό,τι αφορά την δασική, πολιτική. Κοιτώντας το status quo, βλέπουμε ότι έχουμε πιο πολύ ξύλια από ό,τι χρειαζόμαστε και αξιοποιούμε. Θα πρέπει να πείσουμε λοιπόν τους ιδιωτικούς, ε, τους ιδιώτες να σταματήσουν την παραγωγή εν μέρη. Πώς λοιπόν θέλουμε να επεκτείνουμε τις θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό εφόσον δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της ξυλίας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, να υπάρξει συνεργασία ενδεχομένως και με τους ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και νομίζω ότι σημαντικό είναι όλα αυτά να μην τεθούν σε υποχρεωτική βάση, να είναι ναι, θελούσια. <clears throat> να πείσουμε τους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες αλλά και να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δασικών εκτάσεων. Ευχαριστώ. Εξαντλήσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Θα δώσω το λόγο σε εμπειρογνώμονές μας τώρα. Αποφασίστε εσείς ποιος είναι αρμόδιος να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Σημαντικά και χρήσιμα. για τις αλλαγές στην ε, βιομηχανία τη δασική. Στο μέλλον η βιομηχανία θα είναι διαφορετική από ό,τι σήμερα. Αλλάζει συνεχώς. Τα προϊόντα τα οποία θα παράγουμε μετά από 10-20 χρόνια δεν θα είναι τα ίδια για αυτά τα οποία παράγουμε τώρα ή αυτά τα οποία είχαμε την δυνατότητα να παράγουμε πριν από 10-20 χρόνια. Όπως παντού άλλωστε σε όλες τις επιχειρήσεις και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα στον τομέα της ενέργειας είναι η τάση να χρησιμοποιούνται τα ε, απόβλητα της εκμετάλλευσης ε, της δασικής στον τομέα της ενέργειας. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον με τα ευρωπαϊκά δάση και τις δασικές περιοχές. Κοιτάξτε, ε, τα δάση αυξάνονται. Οι δασικές εκτάσεις αυξάνονται και αυτές συνεχώς. Συνεπώς λοιπόν όχι μόνο τα φυτόρια αυξάνονται αλλά αυξάνεται επίσης και η συνολική βασική έκταση. Questions or comments, uh, actually uh, quite many comments or questions uh, they concentrated about differences between. Εν πάση περιπτώσει τώρα για τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια στρατηγική και όχι μια πολιτική. Ε, χρειαζόμαστε εναρμόνιση, χρειαζόμαστε συντονισμό ανάμεσα στις διαφορετικές πολιτικές που να επηρεάζουν σωστά τις διαδικασίες λήψης απόφαση. Αλλά είναι δύσκολο να δει κανεί την ανάγκη που υπάρχει για σωστές πολιτικές αποφάσεις και για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα δάση, ε, ποια είναι τα προϊόντα, πώς θα τα χρησιμοποιούμε. Είναι διαφορετικές οι καταστάσεις στην Μεσόγειο από ό,τι είναι στη Σκανδιναβία. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται να υπάρξει ο συντονισμός αυτός έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχει επίσης και το θέμα του περιβάλλοντος φυσικά και απαιτούνται περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Όταν μιλάμε όμως για θέσεις εργασίας στη βιομηχανία θα πρέπει να δούμε αυτοί οι κανονισμοί, οι περιβαλλοντικοί και η γραφειοκρατία που πηγαίνουν μαζί είναι αυτός ο σκοπός ή μήπως κάποιος άλλος είναι ο σκοπός, πώς θα αποκαταστήσουμε τα δάση και πώς θα εκμεταλλευτούμε ε, τις πρώτες ύλες σωστά. Ε, ε, υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πώς θα μπορέσουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις αναπτύξουμε σωστά. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης στα πλαίσια αυτών των οικοϊπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια στη Βόρεια Ευρώπη όπως είναι και στη Νότια. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Τώρα για τα ορυκτά καύσιμα. Όπως είπα, στη Φιλανδία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Λέμε ότι θα πρέπει να, μέχρι το τέλος του αιώνα θα πρέπει να σταματήσουμε την χρήση πλέον των ορυκτών. Αυτός είναι ο στόχος. Στην Φιλανδία, αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα δάση και αν δεν χρησιμοποιήσουμε το ξύλο, ε, δεν θα τα καταφέρουμε. Πάρα πολύ απλά είναι η μοναδική μας δυνατότητα τα δάση για να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο που έχουμε θέσει. Αν η τακτική που ακολουθούμε μέχρι τώρα είναι η σωστή. Έτσι νομίζω. Νομίζω ότι πράγματι είναι ο σωστός δρόμος για να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ μας και να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση, μια πλήρη στρατηγική και όχι επιμέρους δασικές πολιτικές. Έχω την εντύπωση πάντως ότι το βασικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η εφαρμογή. Νομίζω ότι χρειάζεται σωστή εφαρμογή, ε, συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τους ε, εμπλεκομένους στην δραστηριότητα. Έτσι θα κρυθούν τα μέτρα και οι δράσεις ε, που είναι απαραίτητες. Thank you for the questions. Uh, Mrs. Köstinger raised the issues of... Uh, Η κυρία Köstinger έθεσε τα θέματα της εκπαίδευσης και των προσόντων. Δεν να υπάρχει ευρωπαϊκή μελέτη γι' αυτό, αλλά ξέρουμε ότι πολλά, σε πολλά τέτοια προγράμματα τίθεται το θέμα αυτό. Και να σας υπενθυμίσω ότι σε κάποια προγράμματα υπογραμμίζονται ιδιαίτερως οι νέες ικανότητες που χρειάζονται για την τομέα της βιοοικονομίας και αυτό επηρεάζει και την δασοκομεία και ξέρω ότι σε κάποιες χώρες λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για να αλλάξουν τα μαθητικά προγράμματα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να προσελκυθούν πιο πολλά άτομα, νεαρά άτομα στην δασοκομεία και στις επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για καλές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε διάφορα κράτη-μέλη και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Ο κύριος Έριξον και κάποιοι άλλοι μίλησαν για το θέμα της περιφερειακής διαφοροποίησης. Ναι, σε μία από τι αναφέρθηκα στο θέμα αυτό. η σημασία του δάσους στις διάφορες περιφέρειες θα είναι διαφορετική και στο μέλλον θα υπάρχει ακόμα πιο μεγάλη διαφοροποίηση αναπεριοχή. Η ισορροπία μεταξύ της προστασίας και της παραγωγής θα είναι διαφορετική σε κάθε περιοχή και εξαρτάται λοιπόν από τις αρχές τις αρμόδιες αρχές και από τις περιφέρειες να αποφασίσουν. Θα χρειαζόταν ίσως και θα ήταν ωφέλιμη κάποια, κατεύθυνση. Αλλά αναφέραμε πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά της δασοκομείας στην οικονομία και στην βιοοικονομία. Ο Πολωνός ε, Ευρωβουλευτής ρώτησε και απαντώ. Πήρα τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωστάτ, του Eurostat. Οποιαδήποτε λοιπόν έλλειμμα έχει να κάνει με τον ορισμό που προβλέπει η Eurostat. Υπάρχουν και κάποια πλανεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Μίλησε για κάποια εξ αυτών, αλλά στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν άλλα εναρμονισμένα δεδομένα για το σύνολο της Ευρώπης, προκειμένου να υπάρξει τέτοια σύγκριση. στη συνέχεια σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό κανονισμό και τη ρύθμιση. Αυτό αποτελεί βασικό ζήτημα για τον βασικό κλάδο στην Ευρώπη. Έχουμε το εξής στόχο. Να συμπεριληφθούν οι πολλές διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες σε, ένα, σε μια ομάδα θα πρέπει να ξέρετε ότι σε άλλες ε, περιφέρειες του κόσμου η βασική προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική. Υπάρχει κατακαιρματισμός όπου υπάρχει έντονη βιομηχανοποίηση αφενός και αφατέρου παρθένα δάση τα οποία δεν αγγίζονται. Δεν ακολουθεί αυτό τον, ε, την προσέγγιση η Ευρώπη. Και αυτό συνεπάγεται και διάφορες προκλήσεις και επαναλαμβάνω ότι οι λύσει θα είναι διαφορετικές ανά περιοχή. Αλλά είναι τόσο πολλά τα συμφέροντα, τόσε πολλές και διαφορετικές οι πτυχέ και οι συνιστώσει. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια τεράστια ποικιλία οικονομικών στοιχείων. Αναφέρθηκε και το θέμα των ελαττωμάτων, των ελλημάτων της στρατηγικής. Είναι καλό το ότι περιλαμβάνονται και η βιομηχανική και οι οικονομίες δασικής διαχείρισης. Νομίζω ότι η οικονομική του σημασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω στα θέματα της εφαρμογής της στρατηγικής. Επί της αρχής η στρατηγική πραγματεύεται όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Το βασικό όμως θέμα θα είναι η εφαρμογή και πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία μεταξύ προστασίας και παραγωγής ή μεταξύ οικονομικού και οικολογικού συμφέροντος. Αυτό ε, να απόκειται στις δημόσιες αρχές. Ύστερα. Νομίζω όμως ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. σίγουρα τροφοδοτείτε τη συζήτηση και μας διαφωτίσατε και εμπλουτίσατε τις γνώσεις μας για τα θέματα της, στρατηγικής, της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δάση. Θα παρακαλέσω τώρα τον καθηγητή κύριο Σίσκο να καθίσει για να μας κάνει την παρουσίαση. Minuta przerwy technicznej. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον καθηγητή Σίσκο πρώτα και κατόπιν στον καθηγητή Σάιμονς. Αυτό προβλέπει το πρόγραμμα της ακρόασής μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Όσο ετοιμάζεται ο κύριος Σίσκο, να σας ενημερώσω ότι είναι καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, στις επιστήμες της ζωής. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα δάσκεδαση και πολιτική, διετέλεσε και υπουργό Περιβάλλοντος στην Πολωνία. Αν είστε έτοιμος κύριε καθηγητά, Είμαστε και εμείς έτοιμοι να ακούσουμε την παρουσίασή σας για την αηφόρο διαχείριση των δασών και την πολυλειτουργικότητά τους, προστασία των δασών από τα παράσιτα και από ζυζάνια, αντιπυρική προστασία. Παρακαλώ, κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να πω λίγα λόγια και από πολωνικής πλευράς αλλά και από ευρωπαϊκής απόψεως. Είναι αναφυσβήτητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη χρειάζεται και τα δάση και μια νέα στρατηγική για τα δάση. Αυτό είναι αναφυσβήτητο, αδιαφιλονίκητο. Γιατί, Γιατί έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά ενδιαφέρουν ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ε, έχουμε ε, υποβάθμιση το, των εδαφών, του, των δασών, αύξηση των διεξιδίων του άνθρακα και των καυσαερίων, ε, μεγάλη ανεργία και η καταστροφή υποβάθμιση των δασών ε, επηρεάζει την αύξηση της ανεργίας. Ποιες είναι οι αντιδράσεις. Ε, ε κάποιες νομικές καταρχήν αντιδράσεις στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ε, είχαμε το, το 1992 την ε, έννοια της, ε, της αηφόρου διαχείρισης των δασών. Έχουμε και την σύμβαση πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές, για τη βιοπικιλότητα και τη σύμβαση κατά της απέριμασης. Είχαμε, απερίμωσης. Είχαμε λοιπόν και κάποιες τοπικές αντιδράσεις πέραν των παγκοσμίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το πακέτο ενεργειακών και κλιματικών, το ενεργειακό και πακέτο κλιματικών αλλαγών, της, την σύμβαση για τη βιοπικιλότητα, για το τοπίο. Ε, θα πρέπει να αποτρέψουμε αυτή την υποβάθμιση των δασών και του εδάφους, γιατί έτσι χάνουμε θέσεις απασχόλησης. Πρόκειται για λιλέντε τα θέματα και μπορούμε να πούμε γενικά ότι ε, συνδέονται με συγκεκριμένους ορισμούς και σημαντικά θέματα αιφόρου διαχείριση των δασών και ε, το διοξίδιο του άνθρακα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το οικονομικό ζήτημα που αναφέρεται. Τα χρήματα. Ε, πώς θα εξασφαλίσουμε αυτοχρηματοδότηση αυτών των πολιτικών για να προστατεύσουμε τα δάση και να μειώσουμε και τα καυσαέρια. Λοιπόν, καταρχήν Έχουμε εδώ το, τη διαφάνεια για την απώλεια της βιοπικιλότητας σε μερικές περιοχές της Ευρώπης. Και επίσης το θέμα του άνθρακα, πώς θα το δεσμεύσουμε. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών ταυτόχρονα και έχουμε και κάποιες τιμές, τις, τις τιμές του τόνου διοξιδίου του άνθρακα. Και με βάση τα στοιχεία αυτά ε, ε, που είναι πολλά ε, και κάθε χρόνο αυξάνονται. Ε, ήταν... Ε, και αυτό συνδέεται και με τη βιοπικιλότητα. Είναι 76 τώρα ευρώ ο τόνος. Και έχουμε συσσόρευση του διοξιδίου του άνθρακα πάνω από 450 τόνους και σε αυτό το σύστημα εμπορίας εκπομπών είχαμε πάνω από 10.000 ευρώ κόστος. Και έχουμε και αύξηση του, του διοξιδίου του άνθρακα και, ε, και το θέμα της βιοπικιλότητας που είναι συναφές με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε ένα τέτοιο σύστημα όπου έχουμε πάνω από 160 τόνους ε, ε, άνθρακα και μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα και έχουμε συνεχή, αύξηση και του διοξιδίου του άνθρακα και του άνθρακα. Οπότε ε, είχαμε τις τιμές ε, στο παρελθόν και τις ε, νέες τιμές. Και επίσης έχουμε περιορισμένη βιοπικιλότητα, έχουμε μερικά σπάνια είδη, προστατευόμενα είδη που χρειάζονται συγκεκριμένο σύστημα με παρουσία του άνθρακα στο έδαφος. Επίσης έχουμε φυσικά ε, δάση με τα δικά τους ε, είδη χλωρίδας και πανίδας και αυτό λαμβάνεται υπόψη στο Natura 2000. Έχουμε συγκεκριμένα είδη που μόνο σε ορισμένα σημεία ευδοκιμούν ε, και πουθενά άλλου. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στο σύστημα αξιών μας. Έχουμε πάνω από 300 τόνους άνθρακα και 1000 τόμους διοξιδίου του άνθρακα. Αν τα χάσουμε όλα αυτά, αν αποδεσμευτεί αυτός ο άνθρακας από το έδαφος, από τις καταβόθρες, θα εκλειθεί στο περιβάλλον και θα συμβάλλει στις ε, κλιματικές αλλαγές. Πάνω από 70.000 ευρώ στοιχίζει αυτή η διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Και εδώ έρχομαστε σε ένα σημαντικό θέμα βιοπικιλότητα και οικολογικό. Θα πρέπει υπεύθυνα να με τα δάση και να διασφαλίσουμε τη βιοπικιλότητα και να αξιοποιήσουμε την πρώτη ύλη, την ξυλία, που είναι πολύτιμη. Και ταυτόχρονα μπορούμε να μειώσουμε την πυκνότητα σε διοξίδιο του άνθρακα, χάρη στην αξιοποίηση αυτών των φυσικών καταβοθρών. Βοηθήσω ο πρόεδρος ε, να μιλάω πιο αργά, αλλά μόνο 10 λεπτά έχω, γι' αυτό προσπαθώ να προλάβω να τα πω όλα. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι τα δάση είναι ευκαιρία. Τα δάση και η ανάπτυξη της υπαίθρου. Θα πρέπει λοιπόν να ε, λάβουμε υπόψη και το Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορία Εκπομπών και πώς θα τα συνδέσουμε όλα αυτά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορία Εκπομπών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε υιοθετήσει την οδηγία για, το, για τη δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό. Δεσμεύουμε διοξίδιο του άνθρακα και το αποθηκεύουμε σε βιολογικές περιοχές ε, και έχουμε 60 με 100 ευρώ τον τόνο το κόστος. Ενώ με την σωστή διαχείριση των δασών και με την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας μπορούμε να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τρία μόνο ευρώ κόστος για τον τόνο διοξίδιο του άνθρακα, με τη φυσική δέσμευση του άνθρακα σε αυτές τις καταβόθρες. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε εκατομμύρια ε, στρέμματα και εκτάρια υποβαθμισμένων ε, δασικών εδαφών που θα μπορούσαμε κάλλιστα να τα ανατασώσουμε. γιατί ένα εκτάριο σε ένα εκτάριο μπορούμε 16 τόνους το χρόνο να αποθηκεύουμε εκεί άνθρακα και έχουμε κάποια κονδύλια που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τη βιοπικιλότητα και ταυτόχρονα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιώτο και τη Συμφωνία Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία μόνο θέσεων απασχόλησης στη δασοκομεία. Έχουμε εκατομμύρια εκτάρια υποβαθμισμένων δασών που δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Και αυτά τα δάση μπορούν να απορροφήσουν ε, ε, ακόμη και μισό, 1,5 ε, τόνο, συγγνώμη, διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο. Γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσουμε και αυτά τα υποβαθμισμένα δάση που μπορούν να επιτελέσουν αυτή τη λειτουργία δέσμευση του άνθρακα. Έχουμε και υποβαθμισμένες γεωργικές ακτάσεις, εκατομμύρια. Και επίσης ε, μπορούμε και σε αυτές να έχουμε ένα ε, εκατομμύριο το χρόνο διοξίδιο του άνθρακα δέσμευσης, ε, απορρόφησης στις γέες αυτές, τις υποβαθμισμένες γεωρικές γέες. Έχουμε και κάποιες νομικές πτυχές. Φυσικά πολύ σωστά είπε ένας προλαλήσας ότι κάθε χώρα διαφορετικά διαχειρίζεται τα δάση της. Υπάρχει ένα πολιτιστικό και ιστορικό ζήτημα. Υπάρχει όμως ένα μοντέλο και η Σύμβαση για τις Κλιματικές Αλλαγές και το πρωτόκολλο του Κιώτο λέει ότι όταν απομακρυνθούμε αυτό το μοντέλο και ε, βελτιώσουμε, αυξήσουμε την απορρόφηση θα φτάσουμε σε κάποια όρια. Αυτό το λαμβάνει υπόψη και το πρωτόκολλο του Κιώτο και η Συμφωνία Πλαίσιο των Κλιματικών Αλλαγών. Ποιες τώρα είναι οι επιπλέον δράσεις ε, με βάση τα, τις διάφορες συμφωνίες ε, αναδάσωση, ε, παράταση της ε, ηλικίας ε, υλοτόμησης. Το θέμα είναι να επιτύχουμε η φόρα ανάπτυξη και φτάνουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί αυτό είναι το θέμα της παρουσίασης μου. Θέλουμε να αποφύγουμε την μαζική, μαζική εμφάνιση παρασίτων και ζυζαζίων και φυσικά να περιορίσουμε και τις πυρκαγιές. Αυτό είναι μια επιπλέον δράση. Οπότε από αυτή την άποψη αν δράσουμε και χρηματοδοτήσουμε όλες αυτές τις ενέργειες έχουμε πολλές ευκαιρίες να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των δασών. Και τώρα κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα να τονίσω ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και η Πολωνία το ίδιο. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί τα πολωνικά δάση είναι πρότυπο, παράδειγμα προς μίμηση αηφόρου διαχείρισης δασών παγκοσμίω και στην Ευρώπη. Γιατί εδώ και δεκαετίες ε, ε, υλοτομούμε τα δάση μας, αλλά όλο και αυξάνονται οι δασικές μας εκτάσεις και δεν έχουμε χάσει ε, ούτε ένα είδος χλωρίδας και πανίδας. Και μάλιστα το αντίθετο, απειλούμενα είδη έχουν αυξήσει τους πληθυσμούς τους. Επίσης έχουμε και νομικές διατάξεις και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι η νέα στρατηγική για τα δάση Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνει στόχο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χωρών μελών. Και κατά τη γνώμη μας τα δάση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Και θα πρέπει, όπως λέει και η Σύμβαση για τις κλιματικές αλλαγές, να συνδέσουμε και τα δάση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία Εκπομπών. Γιατί αυτό είναι δίκαιο και θα εξασφαλίσουμε και θα διαφυλάξουμε θέσει απασχόληση και ταυτόχρονα τη βιοπικιλότητα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και να σας προσκαλέσω στην εξέταση των, των εργασιών μας για την απορρόφηση, φυσική απορρόφηση καταβόθρες άνθρακα, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη αξιοποίηση και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα από τα δάση. Σας ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Θα έχουμε στη συνέχεια ευκαιρία να θέσουμε ερωτήσεις ε, κύριε καθηγητά και θα απαντήσετε. Περιμένουμε τα φώτα σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Σάιμονς για να μας παρουσιάσει το δεύτερο θέμα της παγκόσμιες ε, δραστηριότητες για τα δάση και την Παγκόσμια Συμφωνία για τα δάση. Ο κύριος Σάιμονς εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Κέντρο Γεωργοδοσοκομείας που βρίσκεται στην Κένια. Παρακαλώ κύριε Σάιμον, έχετε το λόγο. I'd ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία και την Επιτροπή σας που μας προσκαλέ, με προσκαλέσατε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να σας παρουσιάσω τις απόψει μας για τα δασικά ζητήματα. Θα ήθελα να συζητήσουμε πέντε θέματα τα δάση, βασικά ζητήματα, τις ε, παγκόσμιες διαστάσεις, πώς συνδέονται με την ευρωπαϊκή διάσταση και πώς συνδέονται και με την εθνική διάσταση. Τι είναι λοιπόν το δάσος. Τα δάση αποτελούνται από δέντρα. Ένα δώρο από γενιά σε γενιά ένα από τα λίγα πράγματα που ζουν περισσότερο από τον άνθρωπο. Ο πιο καλός αρχιτέκτονας, ο πιο έξυπνος αρχιτέκτονας, οι πιο ε, καλοί οικοδόμοι ποτέ δεν θα μπορούσαν να καταφέρουν να φτιάξουν ένα δέντρο. Κοιτώντας λοιπόν αυτή την ε, ε καμπή που παίρνουν τα δάση, από την αποδάσωση μέχρι την αναδάσωση, υπάρχει συχνά ένα σημείο όπου ξεχνάμε το εξή. Τα ε, δέντρα αναπτύχθηκαν πριν από 350 εκατομμύρια ε, χρόνια, ενώ τα τροπικά δάση αναπτύχθηκαν πριν από 230 εκατομμύρια χρόνια. Υπήρχε 10 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα. Τα δάση ήταν αυτά που κατέστησαν τον πλανήτη μας ε, ικανό να φιλοξενήσει ζώα και ανθρώπους και επέτρεψαν να ζήσουμε. Ένα από τα προβλήματα με τα δάση είναι το πώς τα ορίζουμε. 18 χρόνια χρειάστηκαν για να οριστεί το δάσος. 8 χρόνια μετά το Κιώτα για να οριστεί ορισμός, να οριστεί το δάσος. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάμε καταρχάς ε, τη θεσμική διάσταση και Κάποιες φορές μιλάμε για την ε, δασική εκμετάλλευση, μιλάμε για ε, δασική έκταση με ή χωρίς δέντρα. Υπάρχουν και δέντρα εκτός ε, δασικής έκτασης. Είναι λοιπόν ένας γρίφος για όλους. Βλέπει κανείς πουθενά σημάδια ενδείξεις αποτάσωσης. Αν θεωρεί ότι μπορεί να δει κάπου σημάδια αποδάσωσης είναι Λάθος, κάνετε λάθος, γιατί αυτή η αποψηλωμένη έκταση είναι μόνο προσωρινό, προσωρινός αποψηλωμένη και αυτό προκαλεί στρεβλώσεις στον ορισμό. Βλέπετε λοιπόν εδώ στη διαφάνεια πώς γίνεται αντρίπτω το δάσος. Τα, όσο πιο σκούρο πράσινο είναι το δάσος, όσο πιο πολύ πυκνή είναι η κάλυψη από δέντρα. Και εδώ βλέπετε ποια είναι η, άποψη των ε, γεωργών για τα τάση. Πώς αντιλαμβάνονται οι γεωργοί τα τάση της κόκκινης κουκίδας και του καθεξής. Πολύ λυπάμαι για το 8% που έχουν χρωματοψία εδώ πέρα στην αίθουσα και δεν βλέπουν το χρώμα από τις κουκίδες. Αλλά έτσι θα πρέπει να βλέπουμε όλοι τα δάση, τα φυσικά δάση και τα τεχνητά δάση από κοινού. Πριν από 20.000 χρόνια είχαμε περίπου 10% ε, κάλυψη δασική. 10.000 χρόνια πριν είχαμε 60% κάλυψη παγκόσμια από δάση και τώρα έχουμε 30%. Έχουμε λοιπόν ε, ε, το ίμιση ή το τριπλάσιο από την δασική έκταση από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Το δάσος λοιπόν δεν θα ε, καλυφθεί από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή στρατηγική, από οποιαδήποτε μεμονωμένη στρατηγική, αλλά σίγουρα θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τα δάση. Α δούμε λοιπόν τι γίνεται σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τα δάση. Τη δεκαετία του 80 στο Νίγηρα, στο Ζίντα, στο νότο τη χώρα, η περιοχή ήταν παραμελημένη και ήταν πολύ χαμηλή η κάλυψη από δέντρα και λόγω της αλλαγής της πολιτικής, μια απλή αλλαγή πολιτικής για την διαχείριση των δέντρων μετατράπηκε σε αυτό που βλέπετε. Και τώρα λοιπόν 5.000 εκτάρια δέντρων, το 3% δηλαδή της δασικής έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει 500.000 τόνους τρόφιμα παραπάνω από ό,τι πριν. Τώρα, να περάσουμε στο δεύτερο θέμα. Ζητήματα που άπτονται των δασών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το νερό, το είδωρο. Πολλά ακούσαμε για τα εμπορικά σχέδια σήμερα το απόγευμα. 200.000 νερό χρειάζεται για να παραχθεί ένα τόνο άνθρακα. 5 ευρώ άνθρακα, το, το κιλό άνθρακα μπορεί να αγοράσετε 400.000 ε, ε, μπουκαλάκια νερό για 5 ευρώ. Καλή τιμή. Δεν νομίζετε ένα σημαντικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα δάση είναι το φόρουμ για τα καταναλωτικά αγαθά, 1-3 ευρώ. Μέχρι το 2020 έχουν δεσμευτεί όλες οι αλυσίδες ε, εφοδιασμού να έχουν 0% αποδάσωση. Αν λοιπόν ρωτιέστε κατά πόσο η Ευρώπη μπορεί να προωθήσει πιο πολλά δέντρα, σίγουρα μπορεί πιο πολλά δάση και σε ό,τι αφορά τους στόχους ε, τους βιώσιμους για το 2030 έχουν να κάνουν με τα δάση 15,4-15,6 και ένα στόχος τους στόχους ε, τους αναπτυξιακούς της Είναι τόσο μεγάλη λοιπόν η διαφοροποίηση των δασών στην Ευρώπη που αναρωτιέστε πώς μπορείτε να τις διαχειριστείτε 250 είδη δέντρων υπάρχουν στην Ευρώπη, 600 στην Αμερική, 1800 στην Κένια. Ε, σε παγκόσμιο επίπεδο 16.000 είδη δασών. Είναι τεράστια λοιπόν η διαφοροποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν περιορίζεται στην Ευρώπη. Τρίτο θέμα. Ε, παγκόσμια διάσταση. Όποια χώρα και να διαλέξετε στον κόσμο, και δείτε την ε, καθαρή αύξηση των δασών. Βλέπετε λοιπόν ότι η Ευρώπη τα πηγαίνει αρκετά καλά. Όπως ε, και... Όχι τόσο καλά όσο η Κίνα, αλλά αρκετά καλά. Μπορούμε ακόμα να βελτιώσουμε όμως την στρατηγική μας. Ξέρετε ποιο είναι το πιο μικρό, η πιο μικρή γραμματεία του ΟΗΕ. Για τα δάση. Τέσσερα άτομα μόνο περιλαμβάνει. Αρμόδια για 4,1 εκατομμύρια εκτάρια δισεκατομμύρια εκτάρια. Δεν ε, δίνουμε τη σημασία που αρμόζει στα δάση. Για την, ε, τα επίπεδα ε, ενίσχυσης για τα δάση έχει, έχουν πέσει. Την τελευταία δεκαετία δραματική αλλαγή. Γιατί τέσσερα ζητήματα αναφέρθηκαν στην, ε, στο Ρίο. Η αλλαγή κλίματος, η απορριμμοποίηση και τα δάση δεν ε, καταλήξαμε σε σύμβαση πλαίσιο για τα δάση. Το 2007 μόλις καταφέραμε και τι καταφέραμε μη δεσμευτικό μέσο, διεθνές μέσο. Και η Ευρώπη έχει ευκαιρία λοιπόν να ηγηθεί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της δασοκομείας. Όχι να χρησιμοποιήσει τη στρατηγική για να ρυθμίσει, αλλά για να προωθήσει, να διευκολύνει την ανάπτυξη πολλά ακούσαμε για τις διεθνείς διαδικασίες στο IPCC, δυστυχώς έχουν διαρρέσει όλο τον κόσμο σε προσαρμογή και απάλυνση. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά ως διαστάσεις. Η γεωργία και η δασοκομεία, ναι, είναι, θέμα, είναι τμήματα του προβλήματος του διοξυδίου του άνθρακα, αλλά και τμήματα της λύσης, ενέργεια, μεταφορές. Δεν πρόκειται να μας ε, σώσουν μόνο αυτά. Και άρα στο διεθνές προσκήνιο υπάρχει μια διεθνής προσέγγιση για την δασοκομεία του χρόνου θα δημοσιευτεί και η ευρωπαϊκή προσέγγιση σίγουρα θα παίξει μεγάλη σημασία. Ας κοιτάξουμε τις ε, ευρωπαϊκές διαστάσεις, τη συνδυασμένη κάλυψη. Να δούμε την Πορτογαλία, 5% δημόσια ιδιοκτησία δασών. Στην Πολωνία 85% το αντίστοιχο ποσοστό. Ένα από τα πράγματα που βλέπουμε λοιπόν στην Ευρώπη είναι το εξή, ότι κατά μέσο όρο υπάρχει χαμηλότερη ε, ιδιοκτησία από τον, από τον δημόσιο κλάδο. Κυρίως είναι σε ιδιωτικά χέρια τα δάση. Το PFC, η πιο μεγάλος οργανισμός πιστοποίησης ε, ε, στις όπως τη Φιλανδία, 100% πιστοποίηση. 11 ε, τέτοιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την παγκόσμια βιοενέργεια και πηγές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δασοκομεία και η βιομάζα θα συμβάλλουν τα μάλα προς την κατεύθυνση αυτή. Κοιτώντας λοιπόν στη Γαλλία, βλέποντας τις ευκαιρίες ακόμα και στις γεωργικές εκτάσεις να αυξηθεί η κάλυψη από δέντρα, όχι μόνο η κάλυψη από δέντρα αλλά και η αποδοτικότητα, η κερδοφορία. Εδώ μπορούμε λοιπόν να έχουμε πιο πολύ ηλετομία, πιο πολύ ξύλο από διάφορες πηγές και ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχουμε χάσει είναι οι μικροί ιδιοκτήτες ε, δασών που θα μπορούσαν να συνενωθούν στους συνεταιρισμού για να χρησιμοποιήσουν, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και για να δημιουργήσουν μεγαλύτερο κέρδος. Και εδώ βλέπουμε ευκαιρίες όχι μόνο για την ξυλία αλλά και για την ανανεώσιμε πηγές ενέργειας. Ευκαιρίες για μεγαλύτερη συλλογή καρπών και προϊόντων ε, από τα δέντρα. Και αυτό προκύπτει από την ε, αναλογία της έκτασης γης. Γιατί το άθροισμα είναι περισσότερα από ότι τα μονομένα στοιχεία και ξέρουμε από το δίκτυο παγκόσμιου αποτυπώματος ότι αυτά θα μας βοηθήσουν στο μέλλον στο παρελθόν ε, μετρούσαμε, προσμετρούσαμε τα πράγματα κάθετα. Στο μέλλον αυτό θα γίνει οριζόντια. Αυτοί που είναι πάνω από τη γραμμή και κάτω από τη γραμμή. Η Φιλανδία, η Βραζιλία και ο Καναδάς ε, έχουν υψηλή κάλυψη από δάση. Αν λοιπόν αυτό είναι το μέλλον στην Ευρώπη και για να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική μας για να προωθήσουμε την βιομάζα, για να διευκολύνουμε τις ιδιωτικές εκτάσεις βασοκομείας ε, προκειμένου να τα πάνε καλύτερα. Γιατί επενδύουμε τόσο λίγα. Οι επενδύσεις στην βιώσιμη διαχείριση δασών και η εφαρμογή της στρατηγικής αποτελούν την πραγματική πρόκληση που έχετε ενώπιον σας και μία σκέψη σας δίνω κλείνοντας. Όσοι προωθούν την βιώσιμη διαχείριση των δασών ζουν περισσότερο, πιο πολλά χρόνια, έχουν πιο πολλούς φίλους, και έχουν και καλύτερη ερωτική ζωή. Και αν δεν μας πιστεύετε, δοκιμάστε και μόνοι σας και θα βρείτε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και τώρα γύρω ερώτα απαντήσεων. Ο κύριος Ντόρφμαν. Αλλά πρώτα η κυρία Κέστιγκερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι δύο αυτές παρεμβάσεις ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, πάρα πολύ καλές. Είχα μία ερώτηση να κάνω για το σύστημα που αναφέρατε και σε ό,τι αφορά την ε, δυνατότητα εφαρμογής. Έχουμε 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ε, δασών στην Ευρώπη. 60% είναι στα χέρια ιδιωτών. Το σύστημα που προτείνεται θα σήμαινε πώληση διαφόρων στοιχείων στο σύστημα. Πώς ε, λοιπόν θα μπορούσε να είναι εφαρμόσιμο ένα τέτοιο σύστημα, πέρα από το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά θα πρέπει έτσι και αλλιώς να μεταρρυθμιστούν στην Ευρώπη. Αυτό είναι ανεξάρτητο. Πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια τέτοια προσέγγιση, γιατί τα αριθμητικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι είναι μη ρεαλιστική η προσέγγιση αυτή. Και για τον κύριο Σάιμονς. Πολύ μου άρεσε η συνολική σας προσέγγιση. Πιστεύω ότι η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η οικονομική αξιοποίηση σημαίνει εμπλουτισμό σε όλους τους τομείς και αυτό σίγουρα θα πρέπει να αποτελέσει στόχο μας στο μέλλον. Έχετε καταπληκτική έκθεση, καταπληκτικό θέμα. Κυρία Πάουλσεν, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν, να σας πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις σας και απευθύνομαι σε όλους τους ομιλητές. Να μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι τα ευρωπαϊκά δάση τελικά είναι απλού τύπου δάση. Έχουμε μια χαμηλή ποικιλότητα εν πολλής ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν λαμβάνουμε πάρα πολύ συχνά υπόψη μας. Στα δάση της Σκανδιναβίας το 99% στην ουσία ανήκουν σε μία κατηγορία. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να, να, να διευκολύνει καλής και άλλα είδη γιατί μόνο το 1% τελικά των ειδών των διαθεσίμων είναι βιώσιμα σε συγκεκριμένες περιοχές. Γι' αυτό και τα δάση μας είναι διαφορετικά από άλλες περιοχές και ιδιαίτερα από τις τροπικές περιοχές όπου εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ειδικά συγκεκριμένα είδη ε, και όχι οικογένειες ειδών όπως ε, σε μας. Είμαστε λοιπόν μια σωστή βάση για μια παραγωγική θα έλεγα ε, υλοτομική δραστηριότητα. Βέβαια αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός, έχουμε δυστυχώς πολύ λιγότερο χώρο για την, ε, ε, για την φύτευση νέων ειδών και γι' αυτό έχουμε και τις πιέσεις της αγοράς, πάντα απαιτούνται όλο και περισσότερα υλικά οικοδομών που προέρχονται από τα δάση, ακόμα και χημικές ουσίες μπορεί να προέλθουν από τα δάση. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι σε 5 με 10 χρόνια από την παραγωγή ε, χαρτοπολτού ε, θα ε, περάσουμε στην παραγωγή υφασμάτων Νομίζω λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα υποπροϊόντα των δασών και για άλλους λόγους όπως ε, την, τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας κτλ. Εγώ ε, ζω στη μέση των Σουηδικών δασών, γύρω μου προς όλες τις κατευθύνσεις έχω μόνο 100, έχω μόνο 100 χιλιόμετρα δάσους, ε, είμαι κυκλωμένη από δάση και γνωρίζω γιατί ομιλώ. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρώτες ύλε από τα δάση, εφόσον τα διαχειριζόμαστε σωστά, είναι ε, τα μόνα άμεσα ανανιώσιμα και περιβαλλοντικά ε, στοιχεία τα οποία μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε τεράστιες ποσότητες αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με προσοχή και να ανανεώνουμε σύνεχώς ε, την, ε, τα προϊόντα τα οποία καταναλώνουμε. Κύριε Σόζουλ, ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, έχω προς σας μια ερώτηση. Μόνο με δύο λόγια, δύο φράσεις μας είπατε για το σύστημα ε, χρηματοδότησης της ε, δοσοκομείας. Μπορείτε να μας αναπτύξετε με περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα αυτό, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, πραγματικά άπειρα στοιχεία. Έχουμε καταρχήν 2% φόρο στο τζίρο από τα δάση Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία οικονομικά για το, την πρότασή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τον ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τη χρήση γης. Γιατί χρειαζόμαστε ε, γη που, για να ικανοποιήσουμε τα, τις επιστηστικές ανάγκες, αλλά αυτή η γη βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιτία των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να μειώσουμε το 40% που έχουμε για να καλλιεργούμε πολύ περισσότερες ε, ε, ε, εκτάσεις και να παράγουμε μόνοι μας τα τρόφιμά μας. Αυτό θα, θα πετήσει περισσότερες γεές, περισσότερα εδάφη. Υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση των βιοκαυσίμων για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Και εδώ συζητούμε για τη δασοκομεία και την ανάγκη να αναδασώσουμε κάποιες εκτάσεις, να φυτέψουμε περισσότερα δέντρα για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερο, ε, μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες. Γιατί το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και άρα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ε, για τη χρήση γης, γιατί βρισκόμαστε σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του κόσμου και φυσικά κλιματικές αλλαγές που θα κλείνουν την πλάστιγα προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Και όλα αυτά τα σενάρια θα, έχουν, ε, επηρεάσουν και την πολεοδομική ε, και αστική ανάπτυξη. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της πόλης των διαφορών μέτρων. Μήπως οι πόλεις μας θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, κάθετα και όχι οριζόντια και θα είναι το μέλλον μας μια ανάπτυξη τύπου Χονγκ και όχι Φλόριδα και ποιες θα είναι οι συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Δασοκομεία από τις επιλογές που θα κάνουμε στην πολεοδομική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βιεγκάς. Okay. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική για τα δάση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή την αίσθηση έχω. Και ευτυχώς θα έλεγα, γιατί στο παρελθόν ε, στην Πορτογαλία εφαρμόστηκαν ε, γεωργικές πολιτικές και σχεδόν ε, εξολοθρεύτηκε η γεωργία. Είχαμε ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, εξολοθρεύτηκε η γεωργία, ευρωπαϊκή αλληλευτική πολιτική και καταστράφηκε ένα μεγάλο τμήμα της Ελίας, ενώ είχαμε παλιά πριν τη ευρωπαϊκή πολιτική πολύ μεγαλύτερη αλληλευτική παραγωγή. Και η δασική πολιτική κοινή τίποτα ε, θετικό δεν προϊονίζεται. Αλλά μία επιβολή εμποροκρατικής άποψης, ε, μερκαντιλιστικής, που ξεκινάει από λύση της αγοράς για να λύσει προβλήματα που μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να λύσει. Το πρόβλημα των δασών σχετίζεται με πολλά άλλα ζητήματα που μας επισήμαναν οι εμπειρογνώμονες και φαίνεται ότι ο κύκλος ζωής είναι πολύ μακρύς, οπότε και από οικονομική άποψη έχουμε μεγάλες δυσκολίες εξαιτία ε, της χρονοβόρας διαδικασίας και υπάρχει και ένας πολύ σοβαρός και μεγάλος κινδύνος για τις χώρες του Νότου. Και επίσης έχουμε μία ε, δομή ε, τα εδάφη μας 3 εκατομμύρια εκτάρια έχουμε έκταση, αλλά 85% όπως είπαμε είναι μικρή, μικρά ιδιωτικά δάση. 400.000 ιδιώτες έχουν δασικές εκτάσεις, αλλά πολύ, μικρή, πολύ μικρές. Και υπάρχει και το θέμα του κτηματολογίου, ε, που ε, δεν έχουμε τέτοιο κτηματολόγιο και έτσι δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια ποιοι είναι αυτοί οι ιδιώτες που έχουν δασικές εκτάσεις και 3% έχουμε μόνο το δασικών εκτάσεών μας ε, σε κρατικά χέρια. Ελάχιστο το δημοσίο δασών. Είναι προφανές για μας ότι μόνο με δημόσιες πολιτικές και με σημαντική ανάμειξη των ε, δημοσίων αρχών θα δώσουμε βιωσιμότητα σε μια πολιτική και θα έχουμε μια πραγματικά υφόρο πολιτική γιατί με το δεδομένο πλαίσιο πολύ δύσκολο θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας, που είναι υπερβολικά φιλόδοξοι. Επίσης πιστεύω ότι τμήμα του προβλήματος ε, οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει το δυναμικό των δασών. Θα πρέπει να προωθήσουμε πολύ περισσότερο τη χρήση του ξύλου να αντιληφθούμε την ανάγκη να αναδείξουμε περισσότερο αυτή την πολύτιμη πρώτη ύλη που είναι το ξύλο. Έτσι θα αποφύγουμε πολλά προβλήματα που έχουμε στην Πορτογαλία. Γιατί πρόκειται για ένα κλάδο που επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή χαρτοπολτού. Και γι' αυτό μετέτρεψε τα δάση μας σε εκτάσεις μονοκαλλιέργειας, κυρίως ευκαλύπτου, μόνο και μόνο για να παράγουμε χαρτοπολτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Βοτσεχόφσκι. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσίαση του κυρίου Σισκό, αν και όλες οι παρουσιάσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Το θέμα της επιρροής των δασών στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι πολύ σημαντικό και ο ρόλος των δασών για τον περιορισμό των καψαερίων, των ρήπων και του διοξιδίου του άνθρακα. Και γιατί υπάρχει πρόβλημα στο να συμπεριλάβουμε τα δάση στον απολογισμό των καυσαερίων και στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Μόνο έτσι με τα δάση θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τα καυσαέρια με την απορρόφηση του διοξιδίου του άνθρακα από τα λάση. Γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην υπολογισμό των δασών, στην εκτίμηση των δασών στις εκπομπές. Γιατί υπάρχει πολιτικό πρόβλημα στο να λάβουμε υπόψη τα δάση σε αυτόν τον απολογισμό. Γιατί έχουμε ολόκληρη συζήτηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη και για τις κλιματικές αλλαγές. Φαίνεται όμως ότι επικρατούν ε, εμπορικά και στεχνιακά συμφέροντα. Και φαίνεται ότι ακριβώς επειδή δεν ε, θεωρούνται οικονομικά προσοδοφόρα τα δάση, τα αφήνουμε εκτός ε, του συστήματος. Αλλά πολύ πιστικά μας είπατε πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα δάση στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ροπέ. Pan Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα τις δύο τελευταίες παρουσιάσεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν πολύ συγκεκριμένες και θα ήθελα να υπογραμμίσω ίσως κάποια θέματα επιπλέον, κάποια θέματα που δεν έχουν ακόμα τεθεί. Στη χώρα μου, τη Λιθουανία, η υλοτομία είναι μια πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα. Μετά από τις επιστροφές γεών στους ιδιώτες, πάρα πολλοί πολίτες α, απέκτησαν δικαιώματα και έχουμε σήμερα πάρα πολλούς ιδιώτες ε, ε, κατόχους με μέσο όρο ε, έκτασης τα 8 εκτάρια. Βέβαια αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στη διαχείριση των δασών και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές σε διάφορες ε, χώρες ε, γύρω από την διαχείριση των δασών, έτσι ώστε να πετύχουμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την απόδοση και να δούμε επίσης και ένα άλλο θέμα που είναι οι αιωλικές ε, τουρμπίνες οι οποίες ε, πολλές φορές τοποθετούνται και σε δασικές περιοχές. Βέβαια στη δική μου χώρα μια τέτοια δραστηριότητα απαγορεύεται. Παρ' όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο ενδιαφέρον και θα ήθελα αν έχετε κάποια γνώμη να μου την ε, εκθέσετε. Σε ορισμένες χώρες επίσης οι σχέσεις ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των δασών, ε, τους, ε, ε, τους κυνηγού, αυτούς που μαζεύουν μανιτάρια, αυτούς που μαζεύουν καρπούς από το έδαφος. Είναι προβλήματα, δημιουργούνται συγκρούσεις και καλό θα είναι να δούμε αν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις δραστηριότητες αυτές καλύτερα. Ευχαριστώ κύριε Σκουσμιόκ. Συνεχίζω τις ερωτήσεις του κυρίου Βοτζεχόφσκι. Έχω ερωτήσεις προς τον καθηγητή Σίσκο. Κύριε καθηγητά, μας αποδείξατε και αριθμητικά πόσο φθηνότερη είναι η απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα από τα δάση από ότι το σύστημα δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Ε, 20-30 φορέ πιο φθηνή είναι η απορρόφηση του διοξίδιου του άνθρακα από τα δάση. Πολύ πιο προσοδοφόρα αυτή η μέθοδο. Και παρόλα αυτά, το θέμα της απορρόφησης του άνθρακα από τα δάση δεν ελήφθη υπόψη στο Σύμφωνο για τις Κλιματικές Αλλαγές. Η συγγήτριά μας, η κυρία Κόστιγκερ, μας μίλησε για αυτό το πρόβλημα της ε, του κατακαιρματισμού της ε, λύσης ε, στην, ε, στην Πολωνία το 85% των δασών βρίσκονται στα χέρια, σε κρατικά χέρια. Είναι δημόσια δάση. Δεν υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός με μικρά δάση σε ιδιωτικά χέρια. Το θέμα όμως της απορρόφησης του διοξιδίου του άνθρακα από τα δάση δεν λαμβάνεται υπόψη στον ε, απολογισμό που γίνεται και στις προσπάθειες για να περιορίσουμε τις εκπομπές καυσαερίων. Μάλιστα, ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των ομιλητών. Έχουμε όμως και εκπρόσωπο από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που είναι εισηγητής ε, της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για το θέμα αυτό, για τη νέα δασική πολιτική. Παρακαλώ λοιπόν τον εκπρόσωπο, δεν ξέρω που κάθεται και αν είναι εδώ. Μάλλον όχι, ας δώσουμε τότε το λόγο στους καλεσμένους μας, στους εμπειρογνώμονές μας για να απαντήσουν. Πολλές ερωτήσεις ε, υποβλήθηκαν. Θα σας δώσουμε αρκετό χρόνο, τουλάχιστον 5 λεπτά στον καθένα για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε πολύ περισσότερες ε, ερωτήσεις από ό,τι χρόνο για να τις απαντήσουμε. Πολύ σημαντικές ήταν όμως οι ερωτήσεις, πολύ εύστοχες. Θα προσπαθήσω να τις ε, συμπυκνώσω στις απαντήσεις. Καταρχήν, ήμουν πρόεδρος της κλιματικές αλλαγές και προετοιμάσει τη διαπραγματευτική θέση σε πολλές συνόδου κορυφή για το περιβάλλον και για το κλίμα. Και θα μπορούσε αυτό ο άνθρωπο, υποφερόμενο, να σα πει το εξή. Το γεγονός ότι το Σύμφωνο για τις Κλιματικές αλλαγέ και το Πρωτόκολλο του Κιώτο αντιμετωπίζουν με ίσο τρόπο δύο δραστηριότητε και τεχνικές, ε, για να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση και να περιοριστούν οι εκπομπές ε, αερίου του θερμοκηπίου και από την άλλη πλευρά για να αξιοποιηθούν ή να αποκατασταθούν ε, κάποιες καταστροφές που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες για να εξασφαλίσουμε καλής ποιότητας είδωρ και αέρα. Και αυτά αυτές οι λύσεις περνάνε από την ε, αναβάθμιση των δασών και των εδαφών και φυσικά με την απορρόφηση του άνθρακα από τα δάση. Γιατί δεν ελήφθη το θέμα της απορρόφησης, ποιος είχε συμφέρον, οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί υπέγραψαν ε, το πρωτόκολλο του Κιώτο και ε, το πακέτο το κλιματικό. Το ενεργειακό όμως πακέτο και το κλιματικό πακέτο δεν έχει καμία σχέση με τη σύμβαση για το κλίμα των Ηνωμένων Εθνών. Ακόμη και αν το διοξείδιο του άνθρακα διαδραμάτιζε πολύ σημαντικότερο ρόλο στις κλιματικές αλλαγές και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πήγμη και δεν έχει μεγάλη επιρροή και δεν έχει αποφασιστική σημασία ε, για, την, ε, ε, το διοξείδιο του άνθρακα. Είμαστε πολύ μικρή ομάδα χωρών. Άλλοι παράγουν πολύ περισσότερες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σημαντικό λοιπόν να πούμε τα πράγματα καθαρά και εξάστερα. Οι εκπομπές ε, αερίων του θερμοκηπίου δεν, ε, δεν την υπόψη ανακράτος, αλλά ανακάτοικο. Και από αυτή την άποψη είναι σημαντικό το πρωτόκολλο του Κιώτο που κάνει ε, διαφορά μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Γιατί είναι 3,5 με 4, τόνου τόνους σε άλλες χώρες, εμείς έχουμε πάνω από 20 και το Λουξεμβούργο 28 τόνους. Και αυτό αφορά μόνο τις ε, εκπομπές αερίου, όχι την κατανάλωση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και τώρα για τα δάση. Ήμουν ε, στις διαπραγματεύσεις ε, και οι 15 χώρες οι αρχικέ Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι θα, θα εγκρίνουν το πρωτόκολλο του Κιώτο υπό έναν και μόνο όρο να μην συμπεριληφθούν τα, ε, τα δάση συγγνώμη, στο σύστημα ε, ανάλυση των εκπομπών. Και έτσι τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιώτο, εξαιρώντας τα δάση από αυτό τον ισολογισμό. Και κυρώθηκε και από τη Ρωσία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο υπό αυτόν τον όρο τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο του Κιώτο. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε γι' αυτό δεν το υπέγραψαν, ενώ είχαν υπογράψει το πρωτόκολλο του Κιώτο και τη, Σύμβαση για τι Κλιματικέ Αλλαγέ, γιατί δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ ε, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα τη ε, απορρόφηση του άνθρακα από τα δάση. Γιατί στην Αμερική έχουν τεράστιες, ε, ε τεράστιες εκτάσεις όπου θα μπορούσαν να, να χρησιμοποιήσουν τις φυσικές καταβόθρες άνθρακα αλλά δεν υπήρξε συμφωνία. Γι' αυτό, γι αυτό και δεν το κύρωσαν το πρωτόκολλο του Κιώτο, παρόλο που το είχαν υπογράψει. Είναι προφανείς αυτές οι αλήθειες για τα δάση. Τώρα, η Πολωνία έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για ε, πολωνική πολιτιστική κληρονομιά. Ανέκαθεν ήταν δημόσια τα δάση στην Πολωνία. Αρχικά ήταν βασιλικά δάση, μετά έγιναν δημόσια κρατικά δάση. Και γι' αυτό δεν είχαμε ιδιωτικά δάση, ελάχιστα ιδιωτικά δάση έχουμε στην Πολωνία. Και τα τελευταία 90 χρόνια τα κρατικά δάση στην Πολωνία είναι 78% του, της συνολικής πολωνικής επικράτειας και με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες για να εξασφαλιστεί η οικολογική ασφάλεια στην Πολωνία. Και όταν λέμε ε, οικολογική ασφάλεια εννοούμε καλ, καλής ποιότητας ε, αέρα, καλής ποιότητας νερό και προστασία της πανίδας, ένα δημοκρατικό κράτος για να το επιτύχει θα πρέπει το 30% της επικράτειάς του να, να καλύπτεται από δάση που θα εξυπηρετούν αυτό το σκοπό της βιοπικιλότητας και της ποιότητας. Αυτό δεν αποκλείει βέβαια, είναι και προσοδοφόρα τα δάση, γιατί στην Πολωνία τα δάση αυτοχρηματοδοτούνται αφενός και αφετέρου επιτελούν όλες τις λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την κοινωνία. Δηλαδή είναι προσιτά στους πολίτες, μπορούν να ε, μαζεύουν μανιτάρια, φράουλες, να κάνουν βόλτες, ακόμη και να κυνηγούν οι Πολωνοί πολίτες. Αυτό προβλέπει το πολωνικό δίκαιο και μάλιστα κατοχυρώνεται το δικαίωμα αυτό και στο Σύνταγμα. Για να εξασφαλιστεί όμως αυτή η ασφάλεια θα πρέπει 30% του, της πολωνικής επικράτειας να καλύπτεται από δάση που θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και ιδιωτικά. Αλλά τα ιδιωτικά δάση έχουν άλλους σκοπούς συνήθως. Γιατί άλλο σκοπού έχουν τα ιδιωτικά δάση, άλλου τα κρατικά δάση, τα δημόσια δάση. Τα δημόσια δάση έχουν στόχο την εξασφάλιση τη προστασία και τη ασφάλεια του πολίτη. Τώρα, γιατί δεν ε, εκμεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτόν τον απλό μηχανισμό. Γιατί δεν έχει πολιτική βούληση. Και επιπλέον, επειδή κάθε χώρα έχει διαφορετική οργάνωση των δασών της και με διαφορετικό τρόπο τα διαχειρίζεται. Τα πολωνικά δημόσια δάση υπόκεινται σε ένα κεντρικό σύστημα ε, με κεντρικό διευθυντή, κεντρική επιτροπή και με μία απόφαση μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρη την πολιτική μας αν χρειάζεται. Εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό, είναι, αυτό προβλέπει το δίκαιο. Γίνονται έρευνες, ανάλυση και αναλαμβάνονται δραστηριότητες. Αυτό έχουμε στην Πολωνία με τα πολωνικά δάση που είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, επαναλαμβάνω. Μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία. Έχουμε συνεργασία με τις ε, τοπικές αυτοδιοικήσεις ε, που, δίνουν, ε, που εξασφαλίζουν πρόσβαση και στους πολίτες, χρηματοδοτούν τα δάση έρευνα, επιστημονικές μελέτες, αλλά και διαφήμιση των δασών, προβολή τους τουριστική. Και αυτό το πολωνικό παράδειγμα θα θέλαμε να το μεταφέρουμε και στην Ευρώπη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Πολωνία είναι παράδειγμα προ μίμηση ό,τι αφορά τη διαχείριση των δασών τη. Έχουμε βέβαια στην Πολωνία και ιδιωτικά δάση. Είναι μικρά βέβαια, είναι μικρές εκτάσεις, κατακαιρματισμένα τα ιδιωτικά δάση και θέλουμε να συνδέσουμε, επαναλαμβάνω, τα δάση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα εμπορία Εκπομπών. Γίνεται αυτό και αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από ε, καταγραφή τους και σε αυτό θα βοηθήσουν τα πολωνικά δημόσια δάση με την εμπειρία που έχουν. Και από αυτή την άποψη είμαστε έτοιμοι ώστε και τα ιδιωτικά δάση και τα δημόσια δάση να τα συνδέσουμε με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μας ενδιαφέρει η διαφύλαξη της βιοπικιλότητας. Στην Ευρώπη έχουμε τεράστια προβλήματα με τη χρηματοδότηση, ακόμη και του Natura 2000. Από πού θα βρούμε τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση. Σας λέω αποκλειστικά και μόνο από την σωστή διαχείριση των δασών, ώστε να εξασφαλίσουμε και την βιοπικιλότητα. Και θα πρέπει να βρούμε τους δείκτες των σωστών ε, των ε, καλών δασών. Ποιος είναι ο βασικός δείκτης του καλού δάσους? Η βιοπικιλότητα. Φυσικά βιοπικιλότητα ανάλογα με το είδος, ε, τον τύπο του δάσους και τις επιτυχίες. Έχουμε μερικά δάση που ε, εξασφαλίζουν και ξυλία και μεγάλη απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά είναι τα δάση με τις καλύτερες επιδόσεις και φυσικά διαφυλάσσουν και τη βιοπικιλότητα. Και χωρίς απώλειες, χωρίς ζημίες, μπορούμε και χωρίς ε, ε, ρήπους να παράγουμε ξυλία, χωρίς ρήπους να παράγουμε βιομάζα από τα κατάλοιπα του, του δάσους και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε τη βιοπικιλότητα. Τα πολωνικά δάση δεν χαρακτηρίζονται από, από σπάνι. Είπατε ότι ε, συνολικά έχουμε 600.000 ε, διαφορετικά δάση. Εγώ είμαι εντομολόγος 2,5 εκατομμύρια διαφορετικά είδη έχουμε παρατηρήσει στα πολωνικά δάση. Μην μου λέτε λοιπόν ότι έχουμε φτωχή βιοπικιλότητα σε καμία περίπτωση. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα δάση για την απορρόφηση του άνθρακα, του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι η φθηνότερη μέθοδος και στο ενεργειακό και κλιματικό πακέτο θα, δεν θα πρέπει μόνο να εξετάζουμε τις νέες τεχνολογίες νέες τεχνολογίες, αλλά το θέμα είναι να δούμε και το χαμηλό κόστος. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμόζουμε τις νέες τεχνολογίες. Γιατί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που δεν είναι οικονομικά προσοδοφόρες. Και το θέμα της ε, αιωλικής ενέργειας. Έχουμε πραγματικά μια μεγάλη άθηση των αιωλικών, της αιωλικής ενέργειας και των ανεμογεννητριών εξαιτία τη πολιτική απόφαση. Ενώ η γεωθερμική ενέργεια είναι πολύ απλούστερη, φθηνότερη και έχει και τεράστιο δυναμικό για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι. Θα ήθελα να σας πω πάντως για τη χρηματοδότηση της δασοκομείας ε, το ανέφερα προηγουμένως, επαναλαμβάνω, αυτοχρηματοδότηση της δασοκομείας στην Πολωνία. Εξασφαλίσαμε αυτή την ανεξαρτησία μετά ε, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα πρέπει, ε, υπήρχε και προεδρικό διάγραμμα, ε, διάταγμα που έλεγε αυτοχρηματοδότηση, εξασφάλιση της αυτοχρηματοδότησης και την προσφορά στην κοινωνία, στο, στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Βέβαια, στην ε, μεσοπολεμική περίοδο είχαμε ένα πρόβλημα στην αυτοχρηματοδότηση και τότε ε, έγινε, έγινε εξαγορά μεγάλων εκτάσεων ιδιωτικών δασών που πέρασαν σε κρατικά χέρια. Γιατί ανέκαθεν η παράδοση της Πολωνίας είναι, ήταν δημόσια δάση και όχι ιδιωτικά. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας κάνω την παρουσίαση και για τη συζήτηση. Η νέα στρατηγική είναι πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε τις ιδιαιτερότητες των χωρών μελών και φυσικά να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουμε αυτές τις ιδιαιτερότητες ώστε να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι το συντομότερο δυνατό μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, διαφύλαξη της βιοπικιλότητας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ήπεθρο, στις αγροτικές ε, ζώνες. Αυτό θα εξυπηρετήσει και την εκτατική γεωργία αλλά και τη βιοπικιλότητα. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητέ. Ε, Λίγο, λίγο κυνηγάτε, γιατί οι γεωργοί μας κάνουν παράπονα ότι εξαιτία των άγριων ζώων χάνουν τις οδηγίες τους. Αυτό είναι όντως τεράστιο πρόβλημα. Στην Πολωνία έχουμε αφρικανική πανόλη των χείρων και είχαμε τέσσερις, τέσσερις θανατώσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κανένα τέτοιο κρούσμα. Και φυσικά θα πρέπει να γίνουν έρευνες και επειδή η μεταφορά είναι ε, δαπανηρή αλλά και οι έρευνες είναι δαπανηρές δεν γίνεται. Πάντως ε, θα πρέπει να αυξηθεί το κυνήγι. Είχαμε τέσσερις θανατώσεις και μάλιστα ε, ε, δεν επιβεβαιώθηκε σε κανένα από αυτά, αυτές τις θανατώσεις κρούσμα τέτοιας επιδημίας της πανόλης της Αφρικανικής. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σάιμονς, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you. Um, Ευχαριστώ πολύ. Οι παρεμβάσεις ήταν περισσότερο σχόλια για την παρέμβασή μου. Τρία πολύ σύντομα σημεία. Πρώτον, έχουμε γέες διαθέσιμες. Ας το χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτό το πλεονέκτημα. Και τα τρόφιμα είναι αρκετά ευθυνά και γι' αυτό ε, πετάμε πάρα πολύ και δεν χρησιμοποιούμε και τα δέντρα με τον πιο έξυπνο τρόπο. Το δεύτερο θέμα ο άνθρακας σαν αγαθό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό το οποίο έχουμε. 15 ε, ευρώ τον τόνο σαν για, ξύλο για καύσιμο και φτάνει στα 100 δις σε εισαγωγικά τον τόνο όταν μιλάμε για τα διαμάντια γιατί και από άνθρακα προέρχονται. Λοιπόν, Τώρα για τον ατμοσφαιρικό άνθρακα θα πρέπει να τεθεί ένα νέο χαμηλότερο όριο. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει σε 2, 3 ή 5 χρόνια. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ ευθυνή η τιμή τώρα. Αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Η Ευρώπη στο τέλος του χρόνου στη Λίμα έχει μια ευκαιρία και στο Παρίσι τον επόμενο χρόνο να αλλάξει την κατάσταση στα πλαίσια των διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιώντας αντιμετωπίσεις χρήσης γης για την υλοτομία, για την γεωργική εκμετάλλευση. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίσκο πάρα πολύ σύντομα παρακαλώ. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για μας. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγουμε πάρα πολλά τρόφιμα. Το, το έδαφος, τα εδάφη που παράγουν θα πρέπει να προστατευθούν από την ε, εξάντληση. Αυτό το οποίο πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε στο έδαφος μια μεγαλύτερη δυνατότητα απορρόφησης και αποθήκευσης άνθρακα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σπάνιο ο Πρόεδρος να μην χρειάζεται να διακόπτει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν χρειάστηκε να το κάνω, να κάνω τον πάρα πολύ αυστηρό. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι έχουμε πλέον ε, την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να ξαναδώσουμε το λόγο στα μέλη. Η κυρία Κώστιγκερ έχει ζητήσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό δείξαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ε, δασοκομεία, τις θέση απασχόληση, τη οικονομική σημασία αλλά κυρίως και του πολύπλευρου ρόλου της βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Και μιας ε, δασοκομείας με μελλοντική διάσταση και τη συνολική σημασία των δασών στην Ευρώπη. Αυτό που προέκυψε στο συμπέρασμα είναι πόσο έντονο περιφερειακό χαρακτήρα έχει το θέμα αυτό. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για το ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι σαφές ότι στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιφερειές μας και το δάσος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο. Ιδιαίτερα η βιώσιμη δασοκομεία είναι κάτι το οποίο απαραίτητο θα πρέπει να κοιτάξουμε σε ό,τι αφορά την στρατηγική για τα δάση και τη σημασία τους. Είναι σαφές ε, το τι συμβαίνει και σε ό,τι αφορά τα δάση που βρίσκονται στα κρατικά χέρια αλλά και στα χέρια ιδιωτών. Και η βιωσιμότητα εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε στην κοινή γνώμη για τη σημασία των δασών από οικολογική άποψη. Το παρουσιάσατε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο και μιλήσατε ότι δεν έχουμε χάσει την ποικιλία των ειδών και των δέντρων στα δάση και φυσικά και από οικονομικής άποψης αν θέλουμε να κοιτάξουμε θέματα ανεξαρτησίας από ορυκτούς πόρους. Είναι πολύ λειτουργικός ο ρόλος των δασών και νομίζω ότι θα πρέπει κοινωνικά να είμαστε περήφανοι για τον πόρο αυτό και να τον αναπτύξουμε στο μέλλον και να μην ξεχάσουμε να λέμε και ευχαριστώ σε όσους ε, διαχειρίζονται τα δάση μας. Είμαι πεπισμένη ότι ο καλύτερος συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι το απαραίτητο. Το χρειαζόμαστε και ήδη έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση της κάποιες σχετικές προσεγγίσεις, θεωρώ ότι μπορούμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω για να βελτιωθούν περαιτέρω τα πράγματα αυτά. Είμαι πεπισμένη απόλυτα ότι ο τομέας της ενέργειας, του κλίματος, του περιβάλλοντος και κυρίως από υπο... άποψη οικονομική είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί λοιπόν ο δασοκομικός κλάδος και να συντονιστεί καλύτερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη σημερινή συνεργασία. Να ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την ε, ζωντανή συμμετοχή, τη συζήτηση, τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Προσβλέπω στην καλή συνεργασία μας τις επόμενες εβδομάδες και θεωρώ ότι η σημασία των δασών και της δασοκομείας ε, προβλήθηκε σωστά σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ καρποφόρα η ακρόασή μας και ευχαριστώ θερμά τους εμπειρογνώμονές μας και τους δύο τελευταίους και τους προηγούμενους. Σας ευχαριστώ όλους θερμά, τα μέλη της Επιτροπής. Λάβαμε πλούσιο υλικό. Θα το επεξεργαστούμε γιατί πραγματικά ήταν πολύ πλούσια η παρουσίαση σε πολλά πλούσια στοιχεία. Αύριο παρακαλώ να είστε παρόντες στις 9 γιατί έχουμε ψηφοφορίες από τις 9. Φέρτε και τις ηλεκτρονικές σας κάρτες ψηφοφορίας παρακαλώ. Και έχουμε και δύο καλεσμένους αύριο για συζήτηση. Παρακαλώ να είστε συνεπείς στην ώρα σας ε, αύριο. Στις 9 θα ξεκινήσουμε. Αύριο δεν θα εφαρμόσω ακαδημαϊκό τέταρτο. Σε 9 ακριβώς θα ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Μην, ξεχνάτε, μην ξεχάσετε τις κάρτες σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.